Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Let me start our meeting. να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Μπορεί να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι εντωμεταξύ. Να ξεκινήσουμε όμως εμείς. Είμαστε στο σημείο 13 της ημερησίας διάταξης της Επιτροπής Ήτρε. συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. TTIP. Opinion. Own initiative. Εξέταση σχεδίου γνωματοδότησης ε, ιδίας πρωτοβουλίας. Όπως γνωρίζετε, η TTIP είναι μια συμφωνία ε, ελευθέρου εμπορίου, την οποία διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Και τα τρία βασικά στοιχεία ε, της TTIP είναι η πρόσβαση στην αγορά, η βελτίωση της ε, εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε ρυθμιστικό επίπεδο και η ε, βελτίωση της συνεργασίας για τον καθαρισμό των διεθνών προτύπων. Αυτά είναι τα τρία πιο ουσιαστικά ζητήματα. Η αγορά, η ε, σε ρυθμιστικό επίπεδο και τα διεθνή πρότυπα. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013. Βρισκόμαστε πλέον λοιπόν 1,5 χρόνο μετά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχουν γίνει 8 γύροι διαπραγματεύσεων και ο επόμενος γύρος θα είναι τον Απρίλιο. Ο τελευταίος γύρος έγινε αρχές Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή ΙΝΤΑ ζήτησε έγκριση για μια έκθεση με τίτλο συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσει για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Επομένως, είναι σημαντικό να ε, υποβάλουμε και εμείς τη γνωμοδότησή μας. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία, ας πούμε σε πέντε λεπτά, την ε, γνωμοδότηση που προτείνω εκ μέρους ε, της Επιτροπής μας και κατόπιν θα ζητήσω από τους ε, σκιώδεις εισηγητές να κάνουν παρεμβάσεις των τριών λεπτών και φυσικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη ε, θα μπορούν να λάβουν το λόγο για ένα με δύο λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις απόψεις της, ε, τα αιτήματά της και τις προτάσεις της. Έχουμε μια ώρα περίπου στη διάθεσή μας, ε, ε, ίσως ε, όχι ακριβώς, 50 λεπτά για τη συζήτηση. Γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός μας εταίρος στην ιστορία της ανθρωπότητας και το πλεόνασμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κοινό μας εμπόριο αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 225 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει πλεόνασμα σε αυτή την περίπτωση. Και οι περισσότεροι συμφωνούν ότι τα συμφέροντα και τα όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μεγαλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι για τις ΗΠΑ από αυτή τη συμφωνία, που σημαίνει ότι περιμένουμε αύξηση 5% και τη χρειαζόμαστε φυσικά αυτή την όθηση, δεδομένου ότι ακόμα ε, βρισκόμαστε σε μια ε, περίοδο στασιμότητας, όχι περίοδο κρίσης, αλλά περίοδο στασιμότητας, κάτι το οποίο βεβαίως είναι επικίνδυνο τα μεγαλύτερα προσκόμματα για το ελεύθερο εμπόριο δεν είναι η τελωνιακοί δασμή και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μάλλον ε, από τους μικρότερους φραγμούς. Ο, ένας από τους μεγαλύτερους φραγμούς είναι ε, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα, πιστοποίηση προϊόντων και τεχνική εναρμόνιση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις και αυτό νομίζω είναι προφανές. Πώς μπορούμε τώρα να αποφύγουμε αυτή την ε, δαπανηρή αλληλοεπικάλυψη, κυρίως στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω το εξής. Η εναλλακτική λύση είναι να δεχτούμε και να εγκρίνουμε τους κανόνες που λαμβάνουμε ε, και που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Κίνα, ε, κανόνες Νοτιού Αμερικής και πρότυπα Νοτιού Αμερικής. Και το ερώτημα είναι κατά πόσον θέλουμε να είμαστε αυτοί που θα καθορίζουμε τα πρότυπα ή απλώς θα δέχονται τα πρότυπα. Ε, ίσως να μην είναι τόσο σημαντικό το γεγονός ότι θα δεχόμαστε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές, αλλά ε, για λόγους υψηλής ασφαλείας θα θέλαμε ε, να μπορούμε να τα διατηρήσουμε αυτά, να έχουμε πρότυπα υψηλής ασφαλείας, ε, ασφάλειας και περιβαλλοντικών προτύπων. Ε, η συνεργασία, κυρίως στην περίπτωση της βιομηχανικής πολιτικής, είναι σημαντική. Σε γενικές γραμμές, Μα ενδιαφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το θέμα της έρευνα και της καινοτομίας. Ε, είναι λίγο, ε, πιο εύκολα τα πράγματα γιατί συνεργαζόμαστε στο, ε, στα προγράμματα πλαίσια εδώ και δεκαετίες με τις ΗΠΑ. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα. Παραδείγματο χάρη το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η ενέργεια. Έχω δύο λεπτά ακόμα, ε, οπότε για το τέλος να σας μιλήσω για την ενέργεια. Θα ήταν πολύ καλό αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να συμπεριλάβει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για την ενέργεια στην TTIP. Ε, νομίζω ότι αυτό ζητάμε και ε, μπορείτε ίσως να το υποστηρίξετε. Κυρίως ελεύθερο εμπόριο καυσίμων και φυσικού αερίου. Τιμές ενέργειας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κατά την άποψή μας και η ενεργειακή ασφάλεια. Θα πρέπει να πούμε ότι οι χαμηλές τιμές ενέργειας στις ΗΠΑ Πολιτείες και οι υψηλές τιμές ενέργειας ε, στην Ευρώπη είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση για τις ενεργοβέρες βιομηχανίες μας, κυρίως για τον τομέα της χημικής βιομηχανίας, το φυσικό αέριο. Ε, σχιστολιθικό φυσικό αέριο επίσης. Ε, από χημική σκοπιά είναι το ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι ε, οι δασμοί για το διοξίδιο του άνθρακα, γιατί έχουμε κάποιες ε, τιμές ε, δασμών για το διοξίδιο του άνθρακα, θα πρέπει να παραμένουν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας TTIP ε, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι τα επίπεδα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα διαφέρουν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Έχουμε ε, τις συζητήσεις που θα γίνουν στο Παρίσι εντός λίγων μηνών και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό και για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι να ξεκινήσουν οι δημόσιες συμβάσεις ε, ε, και να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από πλευράς ΗΠΑ, κάτι που θα μας οδηγήσει σε ανάπτυξη του κλάδου, ε, καινοτομία και είναι πολύ σημαντική και η ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών. Και ίσως και η διαστημική βιομηχανία αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε διότι θα έχουμε αύξηση ε, κατά 6 με 8% εκατέρωθεν ε, για τις δύο πλευρές, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους κοιόδης εισηγητές να παρουσιάσουν και αυτή τις απόψεις τους. Η κυρία Τόγια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες είναι εδώ παρούσα. Εδώ, εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Απλά άλλαξα θέση. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίασή σας. Πολύ περιεκτική, περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά θέματα. Και ευχαριστώ και για το σχέδιο έκθεσης που έχετε προετοιμάσει. Νομίζω ότι εκεί περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, από αυτόν πρέπει να εμβαθύνουμε. Όσον αφορά τώρα τη θέση της δικής μας της ομάδας, εμείς ε, θα κάνουμε σε βάθος δουλειά, θα παρουσιάσουμε, θα καταθέσουμε τροπολογίες, προτάσεις και θέλω κατόπιν να περτώ μόνο σε ορισμένα θέματα. Το TTIP, ε, αυτό το άνοιγμα εμπορικών ανταλλαγών με μια μεγάλη χώρα όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και ε, ανταλλαγή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι ανταλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του εμπορίου που μπορεί να είναι προς όφελος της βιομηχανίας αλλά και της μεταποίησης της δικής μας που εμείς έχουμε καλά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Βεβαίως ε, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή σε αυτή την πραγματικότητα που αφορά ε, ένα μεγάλο κομμάτι της μεταποιητικής σε πολλέ χώρες υπάρχουν αυτέ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό μας ανησυχεί, ότι θα χάσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ανταγωνιστικότητά τους. Άλλε ε, ανησυχίες που έχουμε, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη και σε αυτήν θα κινηθεί η δική μας η πρόταση. Αυτό αφορά την πληροφορική. Εκεί η Ευρώπη προσπαθεί να επικρατήσει. Ε, αυτά σχετίζονται με την πνευματική εργασία και με την τεχνολογία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, ε, κυρίως ε, με την, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν σχέση με την πληροφορική. Όπως είπατε και εσείς, ε, πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο για την ενέργεια και εκεί πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά το κόστος και το όφελος. Το όφελος είναι σαφές, το κόστος σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν πρέπει <clears throat> να χατούμε μέσα από το χαμηλό κόστος της αμερικανικής βιομηχανίας, αλλά να προβάλλουμε τις νέες τεχνολογίες, την πράσινη τεχνολογία και εναλλακτικέ τεχνολογίες, για να μπορούμε και εμείς να προτείνουμε μία σειρά ε, δικών μας προτάσεων. Και τελειώνω με το εξή. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ε, ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές προδιαγραφές, όπως και οι προδιαγραφές της ποιότητας που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Κάτω από αυτό το πρίσμα θα εξετάσουμε εμεί την πρόταση και θα καταθέσουμε τις δικές μας τις ε, τροπολογίες. Εκ μέρου του ECR, των συντηρητικών εκτερνιστών, ο κύριο Μέστερ Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θέλω να σα ε, συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε που προετοιμάσατε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης ε, εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Συμφωνώ με τα γενικά στοιχεία, έχω μόνο λίγες παρατηρήσεις ή αν θέλετε κάποιες ε, προτάσεις ε, που κατά την άποψή μου θα βελτιώσουν το σχέδιο. Στο σημείο υπαριθμών 5 νομίζω είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει... να έχουμε μία μελέτη επιπτώσεων μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή μέτρων για να γνωρίζουμε τις πραγματικές επιπτώσεις. Το δεύτερο, ένα από τα θέματα που συζητήθηκε ευρέως στην Ευρωπαϊκή ε, Προεκλογική Εκστρατεία ήταν να υπάρχει εσωτερική αγορά για ε, ψηφιακά προϊόντα και νομίζω ότι έχει νόημα να τη διευρύνουμε αυτή την αγορά στην περίπτωση βέβαια που καταλήξουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Να συμπεριληφθούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε σε αυτήν την ψηφιακή αγορά. Εγώ λοιπόν ότι πιστεύω ότι έχει νόημα αυτό να αναφέρεται στο, στη δική σας τη γνωμοδότηση. Επίσης, επειδή η Επιτροπή μας εξετάζει τις συγκεκριμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είπε και η προλαλήσασα, είναι σημαντικό να επισημάνουμε το δυναμικό που χαρακτηρίζει αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη βιομηχανία, στην έρευνα, στις τιμές του καταναλωτή, να γίνεται αναφορά σε αυτό έτσι ώστε αυτό να υπάρχει πολύ συγκεκριμένα στην έκθεση. Και τέλος, ε, όσον αφορά στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, νομίζω είναι σημαντικό να ε, τονίσουμε ότι όσον αφορά αυτή τη συμφωνία δεν έχει νόημα να εξετάσουμε το ενεργειακό μείγμα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε εμπόδια ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για την Ευρώπη δεν πρέπει να ορίσουμε εμείς τι είδους πηγές ενέργειας θα χρησιμοποιούν. Είναι σαφές ότι τα πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά. Στην Αμερική έχουν ε, σχεδόν 100% εξαρτησία μέσω του σχιστολιτικού αερίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα είναι πολιτικά ευαίσθητο, πολύ άκρα, άκρα πολιτικά ευαίσθητο ε, και άρα δηλαδή δεν ε, νομίζω ότι αυτός είναι λόγος για να αλλάξει η συμφωνία. Σε γενικές γραμμές, ε, όπως είπατε και εσείς, αυτό είναι ένα από τα ε, λίγα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν για να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ύφεση για να δει φως στο τούνελ και να αποκτήσει μεγαλύτερη ευημερία. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεργαστούμε επικοδομητικά μαζί σας. Τώρα εκ μέρους των φιλελευθέρων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου, ε, αλλά ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ και εγώ για το σχέδιο που συντάξατε, κυρίως για το ύφος που χαρακτηρίζει το σχέδιό σας. Το στηρίζουμε αμερπιφύλακτα. Ε, είναι θετική η συμφωνία TTIP. Εμείς ε, δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα που εκκρεμούν, επί των οποίων πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις που είναι πολύ ευαίσθητα και θέλουμε να επιτευχθεί συμφωνία επ' αυτών. Η συμφωνία όμως TTIP είναι μια ευκαιρία. Ευκαιρία μοναδική στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς λοιπόν σας στηρίζουμε. Τώρα, ένα-δυο πραγματάκια να πω Υπάρχουν πολλά σωστά επιχειρήματα που αναφέρατε και επίσης αναφερθήκατε και στο ότι πρέπει να υπάρχει ισόρροπη προσέγγιση αφενός ε, να δούμε λιγάκι το θέμα των φραγμών στους δασμούς και αφετέρου το θέμα της ευθυγράμμισης ε, κανονισμών. Να πω το εξής, ότι αν τελικά δεν επιτύχουμε ισόρροπη προσέγγιση, αυτό θα παρεμποδίσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Άρα και από αυτού συμφωνούμε απόλυτα. Πρόεδρε, αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο σε κάποιους παραδοσιακούς τομείς που είναι πραγματικά σημαντικοί για τους Ευρωπαίους και θα ήθελα να αναφέρω ορισμένους εξ αυτών η βιομηχανία αυτοματοποιημένων διεργασιών, η μηχανολογία, εκεί συμπεριλαμβάνονται και εξελιγμένα προϊόντα. Και νομίζω πολύ σωστά αναφερθήκατε και στη χημική βιομηχανία και αυτήν πρέπει να την προβάλλουμε. Νομίζω ότι η συνάδελφός μου, Αγγέλικα Νίμπλα, ε, θα μιλήσει για το ενεργειακό μείγμα ε, γι' αυτό εμένα επιτρέψτε μου να κάνω δύο ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Έχουν υποθεί πολλά για τις ε, ΜΜΕ, συμφωνώ και επαυξάνω. Η Αγγέλικα θα πει, νομίζω, ότι πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα. Δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει κάτι που θα το αποκαλούσα συγκαλυμμένος προστατευτισμός στην πραγματικότητα αν εμείς ε, εξάγουμε κάτι θα πρέπει να το έχουμε παράγει εκτός αυτής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι το λέω υπερβολικά. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Τώρα όσον αφορά στις ΜΜΕ, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που θα υποφεληθούν περισσότερο. Πρέπει όμως να δούμε λιγάκι όχι μόνο τους δασμούς αλλά ε, και την ε, πληροφορική, τη συνδυτοποίηση, την πληροφορία γενικότερα. Να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε, θα καταθέσουμε ε, τροπολογίες αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούμε απόλυτα με την κατεύθυνση που δίνεται στο σχέδιό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευπρόσδεκτε θα είναι αυτέ οι τροπολογίε. Κρίμα για τη φωνή σα, γιατί αισθάνομαι ότι πονάτε κιόλα όταν ε, μιλάτε. Ελπίζω να σας περάσει, να σα ευχηθώ περαστικά, ίσω χρειαστεί να μείνετε λίγο άφωνος. Ο συνάδελφο από τους ε, πράσινους. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την έκθεση, θέλω να επισημάνω τέσσερα θέματα, τα οποία κατά την άποψή μας πρέπει να αποκτήσουν εντονότερη διατύπωση. Ενεργειακή Ένωση, ενεργειακή αγορά είναι πολύ σημαντικό θέμα, όπως και αν το πείτε. Κατά την άποψή μας δεν εκπλήσει το ότι το TTIP ε, δεν... Ε, το TTIP ε, θέτει σε μειονεκτική θέση ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ε, Εμά δεν μα αρέσει αυτό το σχιστολιτικό αέριο που υποτίθεται θα εισαχθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα υπονομεύσει ουσιαστικά του στόχου μα ε, για το διοξίδιο του άνθρακα. Θα φαλκιδεύσει την ενεργειακή μας στρατηγική. Το δεύτερο αφορά τη συνεργασία για θέματα κανονισμών. Αυτό θα δείξει ιδιαίτερα την βιομηχανία. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει έτσι ώστε οι δυνατότητες μας για, λήψη αποφάσεων και κανονισμών να μην επηρεαστεί, να μην υπάρξει κανένας είδους περικοπή. Το τρίτο αφορά ε, τις κρατικές προμήθειες το άνοιγμα αυτού του τομέα των δημόσιων διαγωνισμών και κρατικών προμηθειών. Βεβαίως και είναι καλό, αλλά εμείς παρόλα αυτά θέλουμε να διατηρήσουμε τις ε, περιφερειακές ε, προμήθειες, περιφερειακούς διαγωνισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επιμείνει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέβει κάτω από το ισχύον επίπεδο. Και το τέταρτο που είναι εξίσου σημαντικό η ανταλλαγή πληροφοριών, η μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό ε, ωφελεί όλους μας οικονομικά, άρα να βρούμε τους ε, σωστούς κανονισμούς, έχοντας όμως κυρίως κατά νου τα μέτρα εποπτείας ε, που ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Άρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα ε, θα πρέπει να επιμείνει να δημοσιοποιηθούν τα προγράμματα της NSA, να ξέρουμε τι πληροφορίες ε, διοχετεύονται χωρίς τη θέλησή μας πριν τοποθετηθούμε για τις πληροφορίες που επιθυμούμε να δίδουμε και να διαβιβάζουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πούμε εδώ στην Επιτροπή ότι πέραν των δηλώσεων που έγιναν από βορειοαμερικανικής πλευράς υπέρ μιας αλλαγής στην ενεργειακή πολιτική, τα γεγονότα αποδεικνύουν το αντίθετο, ότι είναι υπέρ του φράκινγκ, ότι είναι υπέρ ε, ε, των αγωγών ε, από τον Καναδά που αποτελούν πολύ μεγάλη ζημία για το περιβάλλον αρκεί να δούμε αεροφωτογραφίες για να δείτε τι ακριβώς ε, καταστροφή υπάρχει σε αυτή την περιοχή του κόσμου ή ζουτούν σχιστολιστικό φυσικό αέριο και στρατιωτικά και γεωστρατηγικά μέσα τα οποία ε, μας οδηγούν σε ορυκτά καύσιμα τα οποία είναι ρηπογόνα ε, και περιορισμένα και ολοένα και πιο δαπανηρά διότι ακριβώς ε, για αυτό το λόγο υπάρχουν ε, προσμίξεις και αυτή τη στιγμή αρχίζει ε, να εμφανίζεται το ακριβότερο κομμάτι, το οποίο σημαίνει μεγαλύτερο κόστος όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την κοινωνία. Νομίζω ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε να κάνουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ηγετικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα έπρεπε να αντιταχθούμε σε αυτή την ανεύθυνη ε, ε, στάση στα θέματα των καυσίμων από πλευρά ΗΠΑ και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένε αποφάσει επ' αυτού. Αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα ε, αποφασίζονται μέσω ερώτηση προ του πελίτε, ε, μέσω μια δημοκρατική ένδειξη διαφάνεια, ε, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη όταν ειδικά πρόκειται για το μέλλον μα. Γι' αυτό και ακριβώ είναι διπλά ανεύθυνο και διπλά απαράδεκτο να προσπαθούμε να τροποποιήσουμε το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο ε, δρούμε εμείς, ε, που θεωρούμε ότι θα πρέπει να δρούμε ε, και μάλιστα από την πίσω πόρτα. Ουσιαστικά αυτό προσπαθεί να κάνει η TTIP. Είναι ένας τρόπος να ε, διακυβεύονται οι κυρίαρχες αποφάσεις των Ευρωπαίων πολιτών ε, και οι αποφάσεις για τους φυσικούς μας πόρους, ε, για το περιβάλλον μας, για το μέλλον μας και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το παραγωγικό μας μοντέλο να μην έχουν ληφθεί μέσω των πολιτών μας αλλά μέσω των μεγάλων πολυεθνικών που έχουν αποδείξει πάν φορές ότι τους ενδιαφέρει άποψη της πλειοψηφίας σε δεύτερη μοίρα και όταν δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους ε, θα μπορούν να προσφύγουν και σε ειδικά ε, δικαστήρια διατησίας τα οποία επίσης περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία ώστε τελικά να μπορούν να καταφέρουν να περνάει το δικά τους όταν δεν είναι η πλειοψηφία αυτή που τους υποστηρίζει. Θεωρώ ότι σε ενεργειακό επίπεδο και σε επίπεδο βιωσιμότητας και αφορέ του περιβάλλοντος η συμφωνία TTIP όπως και πολλές άλλες συμφωνίες είναι μια τραγωδία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Κύριο Μπορέλη, από το EFT. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η θέση μας όσον αφορά το TTIP ξεκινάει από μια αντίθεση στην αναφόρον ε, ε, στο ανεφορό άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών και μάλιστα με πρότυπα τα οποία δεν συνάδουν καθόλου με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να συνεισφέρουμε επικοδομητικά στη συζήτηση και να έχουμε μια συνεισφορά η οποία θα προσέχει όσο το δυνατόν περισσότερο του πολίτε, του καταναλωτέ και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ένα από τα βασικά στοιχεία τη γνωμοδότηση αφορά τον τομέα τη ενέργεια. Το τομέα τη ενέργεια η φιλοσοφία μα δεν είναι να υποκαταστήσουμε την εξάρτηση από τη Ρωσία με μια άλλη ασταθή πηγή εξίσου σταθεί όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά να έχουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα ε, βασίζεται στην ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων και στην καταπολέμηση της πατάλης. Ε, να υπάρχει έρευνα στο μέλλον και να, υπάρχουν, να μην υπάρχουν νέες, νέοι διάβλοι προμήθειας ορυκτών καυσίμων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν είναι η Συμφωνία Ελευθέρων Συνταλλαγών ο σημαντικός άξονας που θα μας επιφέρει τις αλλαγές, αλλά η ερευνητική ε, οι μελέτες και οι έρευνες οι οποίες από ό,τι φαίνεται θάβονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το brand fair ε, Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δείχνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εθνικά συμφέροντα, υπερεθνικά σε κάποιες περιπτώσεις και δεν δίνεται συγκεκριμένη σημασία στη ότι έχουν να πούν οι πολίτες. Κατά την άποψή μας η διαβούλευση με την κοινή γνώμη είναι ανεπαρκής. Από τις πρόσφατες διαδηλεύσεις διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει γεωγραφική ισορροπία στη συμμετοχή και τα αποτελέσματα δεν είναι προσωπευτικά μιας ε, περίπλοκης πραγματικότητας των 28 κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια ευπρόσδεκτη μια αξιολόγηση επιπτώσεων, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλα στοιχεία των διαφόρων παικτών, ιδίω όταν συζητούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Uh, And now we go... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στους υπόλοιπους ομιλητές και θα ήθελα να σας ζητήσω οι παρεμβάσει να περιορίζονται στα δύο λεπτά για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Όπως έλεγε... Και ο κύριο Τίτσικα τώρα θα δώσουμε το λόγο στην συνάδελφο πριν την Άλντε που ασχολείται με τα ζητήματα τα ενεργειακά. Πράγματι, υποστηρίζουμε την ε, νομοδότηση όπως την έχετε συγγράψει, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούμε και με την ΙΝΤΑ για να βρεθεί μια ευρεία πλειοψηφία που να υπερψηφίσει ε, αυτή τη γνωμοδότηση και να δώσουμε το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στην Κομισιόν για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Χρειάζεται να είναι ισορροπημένη η γνωμοδότηση στην οποία θα καταλήξουμε και να καλύπτει τα θέματα εκείνα της που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δύο επιτροπών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη στρατηγική, την ενεργειακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργειακή ένωση και τη στρατηγική για την ε, ανεξαρτησία, την ενεργειακή, την προσπάθειά μας να επιτύχουμε αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία με υψηλά πρότυπα και σε φθηνή τιμή. Από αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε το κεφάλαιο το ενεργειακό της TTIP. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για μια διμερή διαπραγμάτευση, επομένω πρέπει να εστιάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, όπω για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή και οι επενδύσει που θα πρέπει να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και να βοηθήσουν τι ε, καινοτομίε για το θέμα αυτό. Όπω επίση υπόθηκε, αποτελεί γλούν οι μικρομεσαίε υποχειρήσει στη ραχοκοκαλιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να φροντίσουμε να μην αποκλειστούν και αντιθέτω να υποστηριχτούν όσο πρέπει. Αυτά είναι τα κυρία ζητήματα κατά την άποψή μου. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Χέκμαρκ. Χόκμαρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ως Πρόεδρος σας ευχαριστώ και ως ε, εισηγητή. Είναι εξαιρετικό το κείμενο που μας υποβάλλεται. Οι τροπολογίες που θα προτείνω θα επιδιώξουν να το ενδυναμώσουν ακόμα παραπάνω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να λεχθεί ότι Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το καλύτερο που μπορεί να επιδιώξει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι να αναθερμάνει τη σχέση της με τις Ηνωμένες Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και χάνει ε, προοδευτικά το ρόλο της Ευρωπαϊκή ε, Ευρώπη ως Ήπειρος Επομένως είναι σημαντικό να δημιουργηθεί αυτή η διατλαντική αυτός ο διατλαντικός οικονομικός χώρος που θα συνδέει τις δύο πιο αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Σε όλα τα πιο σημαντικά ε, ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας συνδέονται με αυτή την προσπάθεια. Η έρευνα, η τεχνολογία, η πληροφορική, η ενέργεια είναι όλοι αυτοί οι τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ τίθεται επίσης το ζήτημα του ανταγωνισμού στην παγκόσμια σκηνή. Υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες σε άλλα μέρη του κόσμου. Διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού. Μπορούν, αν συνεργαστούν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταφέρουν να ανέβουν τα ποιοτικά πρότυπα και έτσι όχι απλώς να έχουμε μεγαλύτερη ε, ανάπτυξη αλλά και πιο ανεπτυγμένη οικονομία ε, ποιοτικά με λιγότερη μόλυνση του περιβάλλοντος, με υψηλότερη ποιότητα. Επομένω, θα έλεγα ότι είναι και προ το συμφέρον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και όλων των κλάδων τη οικονομία με του οποίου ασχολείται αυτή η Επιτροπή να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Και προς αυτή την κατεύθυνση υποβάλλω τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κυρία Χέρστ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Σε επίπεδο αρχής, ε, κανείς δεν έχει αντίρρηση για μια συμφωνία ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Το TTIP όμως δεν είναι μια τέτοια απλή συμφωνία, γιατί έχει κι άλλα, όπως ε, παραδείγματος χάνει τα ρυθμιστικά. Εκεί έχουμε πρόβλημα, γιατί κατ' ουσίαν ε, οι σημαντικές αποφάσεις δεν μπαίνονται σε δημοκρατικό χώρο. Και ποιο μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα επιδεινωθούν οι προδιαγραφές για το περιβάλλον ή για το κλίμα διλήμμα ε, ότι δεν θα ληφθεί μία απόφαση που θα αγνοεί τα κοινοβούλια προς την κατεύθυνση που προανέφερα. Ίσως γιατί αυτό θα είναι οικονομικά αποδοτικό, ίσως διότι μεγάλες ε, επιχειρήσεις ε, μπορούν να καλύψουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που το βρίσκουμε πολύ προβληματικό. Το δεύτερο, η προστασία των επενδυτών. Ε, θεωρώ ότι και αυτή η Επιτροπή πρέπει να εκφράσει με σαφήνεια την άποψή της. Γιατί αν δούμε λιγάκι τους ενεργειακούς ομίλους στη Γερμανία, μιλάμε για 4,7 δις που ε, πρέπει να καταβληθούν. Στην Ισπανία το 8 όταν μπήκε στην κρίση 29 δις ε, ζητήθηκαν από τις ενεργειακές επιχειρήσεις Αργεντινή. 52 περιπτώσεις με τέτοιου είδους αγωγές και πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου που συμβαίνει κάτι παρεμφερές. Διρωτώμε λοιπόν κατά πόσον είναι σωστό αν δεν ε, δημιουργούμε ασφάλεια και ε, καταργούμε αυτή την προστασία των επενδυτών. Όχι να πρέπει οπωσδήποτε ε, να φτιάξουμε ένα όργανο που να είναι και λιγάκι πιο δημοκρατικό. Το τρίτο, ανησυχούμε πολύ όσον αφορά την ενεργειακή αγορά φράκινγκ, ε, ε, πετρέλαιο από πίσα. Ποιος λοιπόν μπορεί να ε, διασφαλιστεί, να διασφαλίσει με ότι θα μπορούν να τηρηθούν οι στόχοι για το κλίμα και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά ας παραμείνουμε λίγο στον ενεργειακό τομέα. Νομίζω ότι εδώ τα πράγματα είναι παντελώς ασαφή και ως εκ τούτου εμείς όσον αφορά αυτό το TTIP όσοι συζητείτε τώρα δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Ε, Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζανανάτο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Συμφωνώ με αυτό που είπατε κι εσείς, ε, στο γεγονός δηλαδή ότι η TTIP ε, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 28 χώρες μέλη μας. Και θεωρώ ότι το αντίθετο θα αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για την Ευρώπη, διότι μεγάλοι ε, οικονομικοί ε, φορείς, άλλες μεγάλες οικονομικές ε, περιοχές θα έχουν ανταλλαγές με τις Ηνωμένε Πολιτείε, και εμείς, η μεγαλύτερη οικονομία της Ιφιλίου, θα έχουμε αποκλειστεί. Από το χρόνο που μου δίνετε θα ήθελα να σας πω μόνο ένα πράγμα για την ενέργεια. Η Ευρώπη εισάγει το 50% των αναγκών της σε ενέργεια για θέρμανση, για μεταφορές, για ηλεκτρική ενέργεια. Το 50%. Και εμείς με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει να εισάγουμε πετρέλαιο, μεθάνιο, φυσικό αέριο και άνθρακα, ιδάλως δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τη βιομηχανία μας. Πόσο θα είναι το μεθάνιο που εισάγουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή θα έχει ανοίξει αυτή η αγορά. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε καθορίσει τις απαραίτητες προδιαγραφές ε, για την ποιότητα της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που θέλουμε να παράξουμε και την ε, ενέργεια που θέλουμε να εξοικονομήσουμε. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Θα αποφασίσουμε εμείς πόσο θα εισάγουμε και αυτή τη στιγμή θα έχουμε αποφασίσει πόσο θα εισάγουμε. Επειδή το σχιστολιστικό φυσικό αέριο είναι μεθάνιο ε, στη χημεία, είναι άνθρακα υδρογόνο 4. Ε, το γεγονός ότι εισάγεται από τη μία ή με την άλλη χώρα εξαρτάται απλώς και μόνο από την τιμή και δεν θα είναι σε καμία περίπτωση περισσότερο από όσο έχουμε αποφασίσει να εκμεταλλευτούμε για τη χρήση που έχουμε καθορίσει προηγουμένως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριο Σταγιάννη. Συμφωνώ με το περιεχόμενο του σχεδίου γνωμοδότησης ε, που μας παρουσιάσατε. Θα ήθελα απλώς ε, να προτείνω δύο προσθήκες. Και για το γενικό τμήμα και για την πτυχή της ε, βιομηχανικής πολιτικής και του τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ενεργοβόροι. Και επίσης όσον αφορά τους δημοσίους ε, διαγωνισμούς, για το γενικό ζήτημα τώρα, τη διαφορά που υπάρχει στις τιμές ενέργειας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλε είναι ένα στοιχείο κλειδί της βιομηχανικής πολιτικής και θεωρώ ότι και σε αυτή τη συμφωνία, ε, την οποία θα πρέπει να προσυπογράψουμε και φυσικά είμαι απόλυτα υπέρ, ε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες ύλε, οι οποίες είναι ουσιαστικές. Η τιμή του φυσικά κυμαίνεται. Αλλά επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μια πολιτική αντίστοιχη με τη δική μας και η ε, μονοπωλιακή σχέση που προσπαθεί ε, να επιβάλλει η Κίνα είναι η ίδια και για τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Θα προσπαθήσω λοιπόν να υποβάλω τροπολογίες για να προσθέσουμε το θέμα των πρώτων υλών. Μια άλλη πηχή που θα ήθελα να τονίσω και για τις ε, δημόσιες προμήθειε και για την πρόσβαση στην αγορά των ε, TIC θα ήθελα να, της πληροφορικής και επικοινωνίας θα ήθελα να σταθώ στην αρχή της αμοιβαιότητας διότι αυτή μας προσφέρει μεγαλύτερες εγγύησεις για τις επιχειρήσεις μας. Εάν δεν υπάρξει άνοιγμα των αγορών ε, και ε, δεν μπορεί να υπάρξει και πρόσβαση εκεί. Εγώ θυμάμαι στην οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες οι τότε επίτροποι Ντεχούχτ και Μπαρνιέ ε, παρουσίασαν ένα κείμενο το οποίο δεν ε, επέτρεπε σε τρίτες χώρες που δεν επέτρεπαν συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών σε δημόσιες προμήθειες να μην μπορούν να συμμετέχουν και αυτές ε, σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Θα προσθέσω λοιπόν και μια τροπολογία, θα σας προτείνω κάτι για να δούμε αν μπορείτε να προσθέσετε και αυτά στην γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρικ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ορισμένε ανησυχίε που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα για δύο σκέλη, δύο πτυχέ τη ε, TTIP. Πρώτον, όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και το δεύτερο είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Αρχικά, για τον ανταγωνισμό. Είπατε ότι η TTIP θα αυξήσει τον ανταγωνισμό, αλλά τελικά το ερώτημα είναι ποιο θα είναι πιο ανταγωνιστικό και γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία του βιομηχανικού κλάδου. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές την μεταφορά των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας σε χώρες ανατολικές, σε χώρες όπου τα μερομίσθια είναι πιο φθηνά. Γιατί να μην υπάρξει με αντίστοιχη κίνηση ε, μεταφοράς δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ, εάν οι συνθήκες εκεί είναι πιο πρόσφορες. Είναι κάτι που συμβαίνει με χημικά εργοστάσια, για παράδειγμα. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ενεργείας στην εδώ πλευρά του Ατλαντικού, στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να μας θορυβήσει. Πρέπει να το εξετάσουμε, να το αναλύσουμε πώς αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει τον κάθε κλάδο ξεχωριστά. Διαφορετικά θα πληγεί ή θα επηρεαστεί τέλο πάντων ο κλάδο τη ενέργεια, διαφορετικά ο κλάδο τη ε, μηχανολογία, των, των ε, εξαρτημάτων των μηχανολογικών κτλ. Περνώ στο δεύτερο θέμα που με απασχολεί, είναι το ζήτημα της πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Το αμερικανικό σύστημα με τις διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις πατέντες, επιτρέπει κινήσεις και προνομική προστασία σε θέματα στα οποία η Ευρώπη έχει επιλέξει να μην δίνει διπλώματα ευρεσιτεχνία. Για παράδειγμα, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στι ε, ευρωπαϊκέ μικρομεσαίε επιχειρήσει. Εάν δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα αυτό μπορεί να δημιουργήσει χάος και να μπλοκάρει τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Ήτρε, κατά την άποψή μου, λέει η κυρία Νάτρη, θα πρέπει να προσθέσει και μια άλλη πτυχή, γιατί ευρωπαϊκές εταιρείες επιδιώκουν να πωλήσουν ε, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ, αλλά τα πρότυπα εκεί είναι διαφορετικά όσον αφορά την ποιότητα ή την ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι και οι δύο πλευρές θα ήθελαν πιστοποίηση υψηλής ποιότητας και ασφάλειας αλλά ίσως επειδή τα πρότυπα αυτά δεν είναι ακριβώς τα ίδια, να δημιουργείται αυξημένο κόστος. Και αυτό πιστεύω πρέπει να αναφερθεί εδώ. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ε, ένα σύστημα ε, δοκιμών των προϊόντων και στις ε, δύο χώρες, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να πιστοποιούνται ως παρκή για τις αγορές και των δύο πλευρών. Και αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο κείμενο που έχει προετοιμάσει ο Πρόεδρος. Συμφωνώ επίσης με τους συναδέλφους που λένε ότι η ενέργεια θα είναι ένα από τα σημαντικά κεφάλαια αυτή τη συζήτηση και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια έξυπνη διατύπωση που να αναφέρεται στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης κάπως να μιλήσουμε για την αρχή, μια, φιλοσοφία αμοιβαιότητα και στην εξέβρεση παρόχων ενέργειας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο περιπλέκει τα πράγματα και στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο. Πάντως θα σας στείλω μια συγκεκριμένη πρόταση διατύπωση αργότερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για αυτό το προσχέδιο γνωμοδότηση. Έχω ένα γενικό σχόλιο πρώτα. Οι διαπραγματεύσει για την TTIP θα έπρεπε να γίνονται σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή δεν ε, γνωρίζουμε την ουσία της διαπραγμάτευσης και δημιουργούνται και διαδίδονται φήμες και αυτό ανησυχεί όλο και περισσότερο τους πολίτες. Ε, έχει ήδη ξεκινήσει μια σύγκριση στους πολίτες μεταξύ της TTIP και της ACTA. Θεωρούν ότι η TTIP, είναι μια νέα ACTA και αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις. Τώρα, η ανάπτυξη της πληροφόρησης των πληροφοριακών συστημάτων σημαίνει ότι θα συλλέγονται όλο και περισσότερα δεδομένα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε μετά να προστατευτούμε από την κατασκοπία, από τις παραβιάσεις της προσωπικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων, όταν έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχει μια τάση να παραβιάζονται αυτά. Και όταν έχουμε διαπιστώσει ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι κάτι που μάλλον περισσότερο ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της, της πνευματικής ιδιοκτησίας, εδώ θα είναι δύσκολο να βρούμε κοινού τόπου, γιατί έχουν μια διαφορετική αντίληψη για το θέμα οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Δελκαστήγιο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με όλους όσους μίλησαν προηγουμένως και θεωρούν ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να υπάρξει απασχόληση, ανάπτυξη και να υπάρξει πρόοδος και ευημερία για τους Ευρωπαίους πολίτες και για, φυσικά και για τους Βορειοαμερικανούς. Πρόκειται για μια ευκαιρία η οποία μας επιτρέπει να έχουμε μια ε, κλιμάκωση από οικονομικής πλευράς που είναι εξαιρετική, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και μεταξύ δύο πολιτικών και οικονομικών περιοχών που συμμερίζονται ε, στην ε, ραχοκοκαλιά των ε, πολιτικών του συστημών τους, στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Πρόκειται λοιπόν για μια μοναδική περίπτωση, όχι λόγω για οικονομικών συνεπειών και φυσικά και κοινωνικών, αλλά και γεωπολιτικών ε, ε, στοιχείων πολύ πιο σημαντικών στον κόσμο που ζούμε πλέον. Γι' αυτό ακριβώ και θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε επαρκώ φιλόδοξοι και ταυτόχρονα πρακτικοί και ρεαλιστέ, προκειμένου να αντιληφθούμε ότι δεν ε, δημιουργούμε ένα καθεστώ ε, ενιαίο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και φτιάχνουμε ένα νέο κράτο έθνο. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα που έχει κράτη έθνη, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ελευθέρου εμπορίου. Πρόκειται για ένα πρώτο στάδιο αυτής της ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Και σε αυτό το πρώτο στάδιο, για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι τα θέματα της ενέργειας, ακόμα και αυτή τη στιγμή, δεν αποτελούν τμήμα της βασικής ε, ε, ουσίας της συνθήκης. Δηλαδή, ακόμα ζητούμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την ενέργεια, για τον τρόπο εφοδιασμού και για τις πρώτες ύλες. Τι να πούμε δε για τον ψηφιακό τομέα που είναι τόσο σημαντικός. Δεν υπάρχει καν ε, κάτι στον ορίζοντα αυτού του σημείου. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε επακριβώς και να επικεντρωθούμε πάρα πολύ καλά σε αυτά που πραγματικά θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτής της συμφωνίας, διότι υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας. Ο χρονικός ορίζοντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάει πέραν ε, της ε, προ... παρούσας Και Επομένως, ε, βρισκόμαστε και εκεί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι πρέπει ε, να φροντίσουμε αυτές οι πτυχές τουλάχιστον, αυτό που σχετίζεται με την ενέργεια και τις πρώτες ύλε να προχωρήσουν, αλλά έχουμε καθυστερήσει ήδη. Εγώ θα ήθελα και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τον ψηφιακό τομέα, αλλά το θέμα είναι ε, Καλό θα, είχαμε, θα ήταν να έχουμε και τους διαπραγματευτέ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά από αυτό τον 8ο γύρο που ολοκληρώθηκε, ποιος είναι ο ορίζοντας που ε, έχουμε ενώπιόν μας και τι ακριβώς ε, θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε από ρεαλιστική σκοπιά και πού θα έπρεπε να επικεντρωθούμε. Ο κόσμος των συμφωνιών ε, ε, ελευθερών εμπορίου με τις ΗΠΑ δεν ολοκληρώνεται με αυτή την έννοια. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι γιατί νομίζω ότι αυτό μας ζητούν μεταξύ άλλων και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ďakujem za som od vás. Εδώ, αν με βλέπετε αριστερά, και εγώ ε, κρίνω θετικά την έκθεσή σας, ε, ε, θετικά κρίνω γενικά τη συμφωνία TTIP. Βεβαίως, Υπάρχει προπαγάνδα, όπως και στη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας, όπου η Ρωσία προηγείται. Και θέλω να σας πω ότι η μία πλευρά δεν δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες, κυρίως όταν τη ζητάνε, ζητάει άλλη πλευρά τις πληροφορίες. Υπάρχουν μελέτες ε, για την αγορά εργασίας, ε, για το περιβάλλον, για την ε, σύντηση, για την ανοτεχνολογία. Αυτό είναι το μόνο όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και σας τα λέω όλα αυτά γιατί επιθυμώ να είμαστε οι καλύτεροι, να έχουμε το πάνω χέρι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτή η συμφωνία μπορεί να μας προσφέρει πωλήσει και θέσεις απασχόληση, αλλά υπάρχουν πολλοί ε, που διαδίδουν ε, ψέματα, ε, όπως σημαίνει και η σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο συνάδελφος κύριος Ρόιλ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, εγώ ζήτησα το λόγο γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή η δυνατότητα να αυξήσει κανείς την αγορά του και με τον τρόπο αυτό να προσφέρει στην Ευρώπη νέες αγορές εργασίας, νομίζω ότι αυτό αφορά τους νέους και τις θέσεις απασχόλησης και όταν υπάρχουν προβλήματα πρέπει να λύνονται τα προβλήματα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί μιλάει κανείς μόνο για προβλήματα. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη. Φαν κλαμπ θα πρέπει να συστηθεί για αυτό το πρόγραμμα και μετά να δούμε πώς μπορούν να λυθούν οι δυσκολίες. Και υπάρχουν θέματα που δεν χρειάζεται καν να λυθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές σε όλους τους τομείς. Ακούω παραδείγματος χάρη ότι ε, λόγω της ε, συμφωνίας αυτής ε, θα επιτρέπεται το φράκινγκ στην Ευρώπη. Μα τις χαζομάρες είναι αυτές, Αναλυσίες. Όποια χώρα στην Ευρώπη θέλει να το κάνει, ήδη σήμερα μπορεί να το κάνει και όλες ε, οι άλλες, ε, αν δεν θέλουν δεν το κάνουν. Αν θέλουν να πάνε να αγοράσουν ε, αέριο από την Ρωσία, με δικό τους πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η γενίκευση των προβλημάτων και να συζητάμε μόνο για αυτά, αυτό το θεωρώ τεράστια δυσκολία σε μια τόσο σημαντική συμφωνία. Να το δούμε αλλιώς, να το πιάσουμε αλλιώς. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία και δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν δυσκολίες δυσκολίες, να δούμε πώς μπορούν να λυθούν οι δυσκολίες αυτές. Αυτός είναι ευφιέστερος τρόπος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρέμβουμε και εμείς σε αυτή τη συζήτηση. Και επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα επειδή πάρα πολλοί βουλευτές αναφέρθηκαν στο χρονικό πλαίσιο για τη συμφωνία, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για την κατάσταση των πραγμάτων. Ως ίσως θα γνωρίζετε, ε, στις 2 Φεβρουαρίου με τον 8ο γύρο διαπραγματεύσεων και ο επόμενος γύρος θα λάβει η χώρα στις 20 Απριλίου, στις Ηνωμένε Πολιτείες αυτή τη φορά. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015 να διεκδικήσουμε πρόοδο υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι ισορροπημένα και μέσα στην εντολή που έχουμε λάβει για διαπραγματεύσεις. Επίσης ελπίζουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε να μπορέσουν να ε, διασφαλίσουν και τη σχετική νομοθεσία κατά τους αμέσους επόμενους μήνες. Και ελπίζουμε αυτό να επιτρέψει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ε, μεταξύ των δύο πλευρών γιατί όπως ξέρετε και οι δύο πλευρές περιμένουν η συμφωνία TTIP να μπει σε καθοριστική φάση. Ο στόχος μας είναι να επιδιώξουμε μια ισόρροπη συμφωνία και βεβαίως ε, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι σήμερα το απόγευμα, αυτό το εκλαμβάνουμε ως μια ευκαιρία. Τώρα, ε, να πω και το εξής, ε, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η δική σας η γνωμοδότηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ε, σε κάποια στοιχεία που και κατά τη δική μας άποψη βέβαια είναι σημαντικά όπως ενέργεια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανικός τομέας, δημόσιοι διαγωνισμοί και επιτρέψτε μου όσον αφορά στην ενέργεια, επειδή τη σχολίασαν πάρα πολλοί βουλευτές, να σας πω ότι προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε ένα ενεργειακό κεφάλαιο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Να απαντήσω και σε αυτά που είπε ο κ. Σταγιάννη σχετικά με τους πόρους. Πράγματι, μιλάμε για την ενέργεια, αλλά μιλάμε για ενέργεια και πρώτες ύλες. Για την ενέργεια λοιπόν είναι σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι δεν αφορά αυτή η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία δεν αφορά στα κυρίαρχα δικαιώματα κρετών να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς τους πόρους. Δεν αφορά στο να αποφασίζει κανείς ε, ή να επιβάλλει κανεί ένα κράτο μέλο στο ενεργειακό μείγμα. Δηλαδή μόλις έχει ληφθεί μια κυρίαρχη απόφαση, στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση των Ευρωπαίων και να μπορούν αυτοί να έχουν πρόσβαση σε εκείνους κάτω από αυτό το πρίσμα αντιμετωπίζουμε τους εμπορικούς περιορισμούς που ενδεχομένως υπάρχουν στις ΗΠΑ για το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Βεβαίως όσον αφορά στην ενέργεια, εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη δική μας τη διαφοροποίηση. Άκουσα ένα μέλος που λέει που ανέφερε ότι δεν θα πρέπει η εξάρτησή μας που υπάρχει με τη, από τη Ρωσία να υπάρχει και από τις ΗΠΑ. Μα κάθε άλλο. Στόχος μας είναι ε, διαφοροποιημένες πηγές έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Και από το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας η ενέργεια είναι πολύ σημαντική. Αναφερθήκατε ε, στο χάσμα στις τιμές που υπάρχει ανάμεσα ε, στις ενεργοβόρες βιομηχανίες από τη μία και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προβλέψεις μας μπορούν να επιλύσουν εν μέρει έστω το πρόβλημα, όχι να το λύσουν πλήρως, γιατί αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και με μία σειρά εσωτερικών αποφάσεων που θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ε, βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, Ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές ε, αναφέρθηκαν και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος μας είναι να μην περιοριστούμε μόνο στα ορυκτά κάψιμα, αλλά να περιλαμβάνουμε και άλλα στοιχεία όπως την ανάπτυξη των ανώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και την ενεργειακή επάρκεια. Πρόεδρε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βεβαίως και είναι η ραχοκοκαλιά της ε, οικονομίας μας αλλά και αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό λοιπόν για πρώτη φορά αποφασίσαμε ε, να διαπραγματευτούμε και ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι καταρχήν οι επιχειρήσεις θα αποκτούν τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που προσφέρονται. Επίσης και για να έχουν μια γενική εικόνα των ε, συμφωνιών και των διατάξεων των συμφωνιών, κυρίως εκείνων που ωφελούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, στο βιομηχανικό τομέα, πολύ σωστά, αρκετοί εξημών επισημάνατε ε, τη βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, χημική βιομηχανία. Αυτή είναι μεταξύ των ε, βιομηχανικών τομέων για τους οποίους επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ένα ειδικό κεφάλαιο στο ρυθμιστικό πλαίσιο της συμφωνίας TTIP. Πρόεδρε, εξάλλου συμφωνούμε με τη σημασία που αποδίδεται στους δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας και πραγματικά βρίσκεται στην ε, πεμπτουσία των ε, διαπραγματεύσεων. Ε, φλεγόμαστε να υπάρχει σωστή πρόσβαση στην αγορά δημόσιων διαγωνισμών των Ηνωμένων να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που έχουν τεθεί από τους Αμερικανούς και τους κείμενους κανονισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ομοσπονδιακό πάντα επίπεδο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εμείς για τις εξηγήσεις σας. Επειδή έχουμε καθυστερήσει όμως λίγο και έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, θα ήθελα να επισημάνω στο τέλος της συζήτησης αυτής ένα-δυο σημαντικά σημεία. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη. Οι περισσότεροι σκιώδεις συζητητές ε, υποστηρίζουν τη γενική γραμμή της γνωμοδότησης. Είμαι εν αναμονή των τροπολογιών σας, θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί συμφωνώ με τις περισσότερες παρατηρήσεις ε, που κάνατε και φυσικά και από τα ε, άλλα μέλη τα όσα ακούστηκαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Καλωσορίζουμε και τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, τον κύριο Λάγκε, ο οποίος είναι αρμόδιος και για το TTIP. Ε, να σας πω ότι δεν δημιουργούμε ένα νέο κράτος έθνος, όπως είπε η κυρία αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι απλώς διαπραγματευόμαστε το άνοιγμα της αγοράς για εμπόριο. Υπάρχουν αντίστοιχε σχέσει αυτή τη στιγμή με την Ιαπωνία ή την Νότια Κορέα. Γνωρίζω ότι δεν είναι ακριβώ το ίδιο ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία, αλλά η συμφωνία λειτουργεί αρκετά καλά. Επομένω, τα πάντα εξαρτώνται από τι διαπραγματεύσει. Εσεί αναφέρεστε σε διαφάνεια, πλήρη διαφάνεια. Ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ε, ε, ζωντανή ε, μετάδοση μέσω διαδικτύου των γύρων διαπραγματεύσεων και πλήρης περιφερειακές εκθέσεις στο διαδίκτυο. Είναι απαραίτητο να τις διαβάζουμε όλες αυτές φυσικά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας. Η δική μας ευθύνη είναι να ξεκινήσουν οι συζητήσεις στην περιοχή μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν τέλει εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν, διότι ήταν το δραματικό ερώτημα που μας απασχολούσε. Ποιος ε, θα μας εγγυηθεί τα πάντα, είπε η κυρία Έρνστε, οι διαπραγματευτέ μας, μας και εν τέλει εμείς που είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ψηφίσουμε επί του ζητήματος και θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως τις συζητήσεις μας με τους πολίτες. Κάποιοι συνάδελφοι, ο κύριο Ρόιλ, ο κύριο Μάνκα, ο κύριο Τζανονάτο, ουσιαστικά ε, απάντησαν ε, στους συναδέλφους που εξέφρασαν τι αμφιβολίε μα. Οι αμφιβολίε είναι προφανεί. αλλά ε, πρέπει να σα πω ότι ε, κάποιοι συνάδελφοι ε, δεν ήσασταν παρόντες. Ε, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που διαμαρτυρήθηκαν αρκετά. Ο κύριο Ετσενίκε είχε πρόβλημα εν γέννη με το γενικότερο ζήτημα δεν θα θέλαμε να υπάρξει κανενό είδους κοινωνικό ή περιβαλλοντικό dumping. Αυτό είναι προφανές, αλλά εξαρτάται και από τις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να είναι ανοιχτέ, ισχυρέ διαπραγματεύσει. Τα πάντα είναι μπροστά μα. Και ε, για μα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένω, ε, δεν θα αρκεί απλώ να διαμαρτυρόμαστε θα πρέπει να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις. Πλήρη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα, για παράδειγμα. Σίγουρα θέλουμε να ανοίξουμε τις αγορές μας, γιατί περιμένουμε φθηνότερη ενέργεια στην Ευρώπη και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Α, να απαντήσω στον κύριο Γκέρεκ, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται και από τις τιμές της ενέργειας. Θα δούμε πώς ε, θα έχουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα είναι πολύ δύσκολο. Πολύ σωστά είπε η κυρία Ομπάτσκα. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι το θέμα των δημοσίων συμβάσεων σίγουρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, με την παρούσα κατάσταση. Οι δημόσιες συμβάσεις στις ΗΠΑ είναι κλειστές για τις επιχειρήσεις μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Σίγουρα έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, σίγουρα θα γίνουν πολλοί γύροι συζητήσεων και ε, δικαίως κάποιοι είπαν ότι από αμερικανική σκοπιά υπάρχει μία προθεσμία για το τέλος του 2016, γιατί θα ήθελα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος της θητείας Ομπάμα. Ε, ευτυχώς η δική μας η προθεσμία είναι το 2019, γιατί τότε λίγη η δική μας η θητεία, εμείς έχουμε πιο πολύ χρόνο. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε στις διαπραγματεύσεις γιατί θα μπορεί ε, να μας βοηθήσει. Το να υπάρξει άνοιγμα στις αμερικανικές αγορές θα μας βοηθήσει. Αλλά δεν θα πρέπει να διαπραγματευτούμε ε, βιαστικά. Πρέπει να δούμε τα πάντα σημείο προς σημείο και στο τέλος είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει μεγάλη επιτυχία και για τις δύο πλευρές, και για τις ΗΠΑ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω την άποψή σας, καθώς επίσης και όλες τις αμφιβολίες και ε, το γεγονός ότι για κάποια σημεία δεν μπορείτε να συμφωνήσετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τους διαπραγματευτές μας. Η γνωμοδότηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. 27 Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα, διορία για την κατάθεση τροπολογιών. Τα πάντα λοιπόν εντός της εβδομάδας. 27 του μηνός, 12 η ώρα. Παρακαλώ να στείλετε τις τροπολογίες σας. Είναι πολύ χρήσιμες, πολύ σημαντικές για το σχέδιο γνωμοδότησης. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου τώρα να καλέσω εδώ τους πέντε ομιλητές για την ακρόασή μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, συζητήσει για το TTIP σήμερα. Το επόμενο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 14, είναι η συζήτηση για το TTIP και πρέπει να σας πω Ίσως θα πρέπει να πω για το σημείο 16, γιατί μάλλον δεν θα μείνουν οι περισσότεροι μέχρι τις 6.30. Η επόμενη συνεδρίαση ε, της Επιτροπής Ήτρε είναι στις 23 ε, Μαρτίου του 2015, 3 με 6.30 και 24 Μαρτίου, 9 με 12.30 και 3 με 6.30. 23 και 24 Μαρτίου λοιπόν είναι η επόμενη συνεδρίασή μας και τώρα να περάσουμε στην ακρόαση για τις συνέπειες της ε, TTIP στους τομείς πολιτικές της ε, Επιτροπής ΙΤΡΕ. Να καλωσορίσουμε τους πέντε ομιλητές μας, τους προσκεκλημένους μας και φυσικά τον συνάδελφο από την Επιτροπή ΙΝΤΑ, πρόεδρο της Επιτροπής ΙΝΤΑ, τον κύριο Μπέρντ Λάγκε. Να πω δύο λόγια στην αρχή της συνεδρίασής μας Well, I've got so many mm, sheets uh, and documentation. Έχω πολλά ε, έγγραφα εδώ μπροστά μου και πρέπει να βρω το σωστό. Σημειώσει του Προέδρου, δεν είναι αυτό. Α, να το, να το. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτηση για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε για την TTIP και θα θυμάστε πολύ καλά όλα τα αποτελέσματα και το πόσο φλέγον είναι αυτό το ζήτημα και η συζήτηση ε, αυτή προσφάτως σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυξανόμενη αντίσταση στην TTIP και θα πρέπει ε, να το γνωρίζουμε αυτό εάν πιστεύουμε πραγματικά στις διαπραγματεύσεις για την TTIP και στο άνοιγμα των αγορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ε, πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και να αναλάβουν και την ευθύνη γι' αυτό. Κάθε συζήτηση είναι όλο και πιο φλέγουσα. Και είναι περισσότερο ιδεολογία η συζήτηση παρά απτά γεγονότα. Δεν αρέσει στον κόσμο να βλέπει το διαδίκτυο, να βλέπει τις διαπραγματεύσεις και να ακούει τις εκθέσεις, ε, απλώς και μόνο ε, γιατί είναι ιδεολογικά αντίθετη σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την TTIP. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, να αλλάξει η ιδεολογική αντίσταση και να ε, περάσουμε σε μια ε, πραγματική συζήτηση. Αυτό είναι το βασικό καθήκον, ο βασικό στόχος αυτής της ακρόασης. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου, ε, εν είδη έναρξης, να ζητήσω τώρα το λόγο, να δώσω συγγνώμη τώρα το λόγο στον συνάδελφο από την Ίντα για να κάνει μια σύντομη δήλωση, πολύ σύντομη γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο, Μπέρντ. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο για τι παρατηρήσει σας. Σα ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Θα έλεγα ότι αυτή η ακρόαση γίνεται σε μια χρονική στιγμή κατάλληλη, επίκαιρη. Υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις, παρερμηνίες. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και στην Επιτροπή Ίντα και είχε έρθει η στιγμή να κάνουμε τον απολογισμό των διαπραγματεύσεων τον τελευταίο 1,5 χρόνο και διαμορφώνοντας τη θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τις νέες κατευθύνσεις στους διαπραγματευτές. Προσωπικά είμαι πλήρως φοβισμένος ότι η TTIP θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Ευρώπης και το στόχο που έχουμε θέσει για το 20% του ΑΕΠ στο 2020. Αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε σε όλους τους ε, τομείς της πολιτικής μας είτε είναι ζητήματα αρμοδιότητας της ε, Επιτροπής Έρευνας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ή της ΣΥΝΤΑ, του Διεθνούς Εμπορίου ή άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου που συνολικά είναι 14 στον αριθμό οι επιτροπές του Κοινοβουλίου που έχουν να συνεισφέρουν μια γνωμοδότηση, να εκφράσουν μια θέση πάνω στις διαπραγματεύσεις για την TTIP και αυτό είναι κάτι μοναδικό στα χρονικά του Κοινοβουλίου. Χωρίς αμφιβολία, η ενέργεια, η βιομηχανία, η ενεργειακή ασφάλεια, τα τεχνολογικά πρότυπα ποιότητας, είναι σημαντικά θέματα και ταυτόχρονα ε, είναι κάτι που μας αφορά όλους, πρέπει να νομίζω όλοι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να υπάρχει ένα ξεκάθαρο, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις διαπραγματεύσεις για την TTIP, πώς θα συνδυαστεί η συμφωνία αυτή με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, πώς θα υπάρχει αμοιβαιότητα στην αναγνώριση των προτύπων που να διευκολύνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτή την αρχή που έχουμε διατυπώσει, που είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις μικρές εταιρείες, τις μικρές επιχειρήσεις πρώτα ευχαριστώ. Από την πλευρά μου θέλω να ακούσω τους ειδικού. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Το πρώτο μέρος της ακρόασης ε, θα το συντονίσω ο, ίδιος και το δεύτερο μέρος ο συνάδελφος από την ΙΝΤΑ. 14 γνωμοδοτήσεις. Και το ερώτημα είναι προς εσάς. Είστε διατεθειμένοι να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τη γνωμοδότηση της ΙΤΡΕ. Απάντηση είναι βέβαια. Ο πρόεδρο ε, τη Ήτρα διακόπτει. Ναι, εντάξει, ωραία, αφού είπατε ναι, βεβαίω, ε, εγώ, εγώ καλύφθηκα αυτό. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα άλλο. Απλώ δεν θέλω να, ακούσω το κομμάτι τη φράση που ξεκινάει με το ναι, αλλά. Οκ. Okay. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Νόβακ. Ο Λεχνόβιτ, με συγχωρείτε. Ε, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εταιρική Σχέση για την Ενέργεια στην Κεντρική Ευρώπη. 4, για 14 λεπτά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ιδιαίτερα ευτυχής που έχω τη δυνατότητα να απευθυνθώ στις δύο αυτές τις του Κοινοβουλίου για ένα ζήτημα τόσο σημαντικό, τόσο ενδιαφέρον. Εκτός μικροφώνου μιλήτη. Σα συγγνώμη. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ ένα κονσόρτιουμ ε, οργανισμών και ε, ε, φορέων που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Θάλασσα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της TTIP. Η TTIP θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει την αύξηση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θέσεων εργασία. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις διάφορες, ε, στους διάφορους οικονομικούς κλάδους στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να αντιληφθεί ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες προβλημάτων που συνδέονται με την TTIP. Η πρώτη κατηγορία έχει σχέση με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και η δεύτερη κατηγορία προβλημάτων είναι εσωτερική. Είναι τα προβλήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και κανέναν άλλον. Το ρυθμιστικό της πλαίσιο, για παράδειγμα. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση ε, στο αργό πετρέλαιο και στις ενεργειακές πηγές γενικότερα, έτσι ώστε να έχει ενεργειακή αυτονομία, ενεργειακή ασφάλεια η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σήμερα η χημική βιομηχανία στις ΗΠΑ αναπτύσσεται ε, ραγδαία εξαιτία ακριβώ αυτών των χαμηλών τιμών στην ενέργεια. Στον χάρτη που βλέπετε αυτή τη στιγμή στη, διαφάνεια που προβάλλεται στην οθόνη, ε, οι βιομηχανίες στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επενδύσει στον τομέα του αζότου το 43% του κύκλου εργασιών τους, ενώ ε, παράλληλα έχει αυξηθεί η ανεργία στις ΗΠΑ. Αυτό το λέω γιατί αυτές οι νέες πηγές ενέργειας, ε, μάλλον οι χαμηλότερες τιμές, ε, το χαμηλότερο κόστος της ενέργειας στις ΗΠΑ ε, εξηγείται κυρίως εξαιτία της χαμηλότερης φορολόγησης και όχι μόνο και όχι κυρίως εξαιτία των νέων και διαφοροποιημένων πηγών. Στον τομέα λοιπόν της χημικής βιομηχανίας έχουμε 6,5% δεσμούς για να προστατεύεται η αγορά των χημικών προϊόντων, ε, προϊόντων ε, επεξεργασίας. Μέσα σε 5-10 χρόνια αυτή η δασμή, αυτή το, το κόστος πρέπει να εξαλειφθεί για τη χημική βιομηχανία. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας 10 χρόνια Σύμφωνα με την ρήτρε που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών θα έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι δασμοί να αυξηθούν από τη μία πλευρά εφόσον ε, εξηγηθεί στον εταίρο, στον, στην άλλη πλευρά γιατί γίνεται αυτό. Καλωσορίζουμε τι πληροφορίε που μας έδωσε η Γενική Διεύθυνση Ενία Αγοράς και επιχειρηματικότητα, και σύμφωνα με τι οποίε ο κανονισμός REACH δεν πρόκειται να υπονομευθεί, δεν πρόκειται να, να, εξαιρεθεί και οι ε, ε, επιχειρήσεις των ΗΠΑ θα είναι υποχρεωμένες να καταχωρούνται και αυτές στο σύστημα REACH. Ένα άλλο ζήτημα σημαντικό που είχε ανακύψει στη διαπραγματεύση τον τελευταίο καιρό, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την οικονομία που συνδέεται άμεσα με την τελική τιμή καταναλωτή των προϊόντων. Δείτε τα στοιχεία για το 2013. Οι κατακεφαλήν εκπομπές το 2013 ανέρχονταν σε 16,55 χιλιόγραμμα ανά άτομο, ενώ στην Ευρώπη ήταν 7,35. Αυτό δείχνει ότι το κόστος παραγωγής στις ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τίθεται το ερώτημα πώς εξηγείται αυτή η διαφορά. Υπάρχουν διαφορές φυσικά στην προσεγγίση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για τη μείωση των εκπομπών. Και βλέπετε ότι τα αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα προσπάθειες μείωσης αυτών των εκπομπών δεν είναι ακόμα ικανοποιητικά. Εσωτερική νομοθεσία. Η CEP e υποστηρίζει τις ε, συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο πλαίσιο του TTIP, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ασφαλές πλαίσιο ρυθμιστικό που να ευνοεί τον ανταγωνισμό και έτσι να ε, δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας. Στις ενεργοβόρες βιομηχανίες θα πρέπει να καταφορηθούν αυτές σε ένα ειδικό κατάλογο έως το 2020 και μετά το 2030 να ακολουθήσουν την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για να μειώσουν τις εκπομπές τους, ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Επισημαίνω όμως ότι ορισμένες από αυτές τις ε, επιχειρήσεις, από αυτές τις βιομηχανίες οι οποίες είναι στην η παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βελτιώσουμε την, ενεργειακή, την αποδοτικότητα μάλλον των, ε, της παραγωγής ενέργειας. Και τέλος, οι βιομηχανίες οι οποίες εκπροσωπώ θα έλεγα ότι δεν αντιμετωπίζουν ευνοϊκές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο ευνοϊκές μάλλον όσο αυτές που αντιμετωπίζουν στη ΣΥΠΑ. Εμείς θα θέλαμε όμως να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας εδώ, στην Ευρώπη, και πιστεύουμε ότι η TTIP μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Σας ζητώ λοιπόν να λάβετε υπόψη σας ξεχωριστά την ειδική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες οι οποίες πρέπει να αναβαθμίσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα να εφαρμόσουν το σύστημα NSA. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Όλεχνόβιτς. Κύριε Στεγιάντε, δεύτερος ομιλητής. Έχετε λόγο. Και εσείς για 10 λεπτά παρακαλώ.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 Γεια σα. Κατάγομαι από την Ισπανία. Είμαι από ένα οικολογικό κίνημα που λέγεται Οικολόγια εν δράση και ότι κάποιες από τι διαφάνειες, επειδή έχουμε μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μα και πολλέ από τι διαφάνειες που θα δούμε θα χρειάζονταν πολύ περισσότερο χρόνο για να τι εξηγήσουμε καλύτερα, θα τι πω λίγο συνοπτικά και επομένω από εκεί και πέρα για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε υπάρχει η διεύθυνση ηλεκτρονική ταχυδρομείου μου στο τέλο και με φυσικά και στη διάθεσή σα. Να ξεκινήσω με την παρουσίαση. Καταρχάς, Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία που από ό,τι άκουσα από την προηγούμενη συζήτηση νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστά. Καταρχάς να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται κατά 50% σε θέματα ενέργειας από τρίτες χώρες και θα πρέπει να δούμε ότι καταρχάς ε, για τα ορυκτά καύσιμα ε, στο πετρέλαιο εξαρτώμαστε κατά 85% και στο φυσικό αέριο κατά 60%. Ακούγοντας φυσικά τις προηγούμενες συζητήσεις ε, νομίζω ότι είναι ανησυχία όλων αυτό. Επιπλέον να τονίσω ότι αυτή η ενεργειακή κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κυρίως αφορά τις μεταφορές. Οι μεταφορές είναι πάνω από το 30% της πρωτογενούς ενέργειας και είναι ένας πολύ ευάλωτος τομέας διότι εξαρτάται πρωτίστως από το πετρέλαιο το οποίο αναφέραμε ότι ελάχιστα ελάχιστο ε, λαμβάνουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πλαίσιο σημαίνει ότι είναι ευάλωτη η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά, κυρίως ε, στα όσα προέκυψαν το 2008, το οποίο νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι, ε, η οικονομική κρίση, μια χρηματοπιστωτική κρίση και αυτή τη στιγμή ζούμε μια στιγμή παγκόσμιας αλλαγής, αλλά υπάρχουν και γεωπολιτικές αλλαγές, όχι μόνο σε ενεργειακό επίπεδο, υπάρχει ε, μη αναστρέψιμη υποβάθμιση της γης, ε, υπάρχει κλιματική αλλαγή και ζούμε μια περίοδο αλλαγής. Επομένως υπάρχουν δύο δρόμοι ουσιαστικά, ιδίω όταν υπάρχει ένα πλαίσιο αλλαγής και αυτό είναι δύο διαφορετικές στρατηγικές. Υπάρχει η στρατηγική του business as usual, δηλαδή να συνεχίσουμε όπως κάνουμε, αυτό που, συνεχίζουμε, που ξέρουμε να κάνουμε και ο άλλος τρόπος είναι να προσαρμοστούμε, να προσαρμοστούμε στις υφιστάμενες συνθήκες και στις αλλαγές που προκύπτουν. Ε, προφανώς το να συνεχίσουμε με αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι το πιο εύκολο, να συνεχίσουμε με την αδράνεια που έχουμε μάθει, διότι το να αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε στο νέο πλαίσιο ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια βεβαιότητα και να αλλάξει η κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή, που πάντα σημαίνει ότι θα πρέπει λίγο να ξεβολευτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να συνεχίσει ε, με αυτό το business as usual, ε, δεν αντιλαμβανόμαστε κάποια αλλαγή, γιατί η αλλαγή σημαίνει ότι θα αλλάξει και το μοντέλο ενέργειας της κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει, να προσπαθεί να αποκτήσει τους ενεργειακούς πόρους που δεν έχει στα εδάφη της από άλλες χώρες, να τις λάβει από αλλό και επομένως ε, ε, διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση σημαίνει να προσπαθήσει να εξαρτάται λίγο λιγότερο από τη Ρωσία και να εξαρτάται περισσότερο από χώρες όπως οι ΗΠΑ ο Καναδάς. Χώρες που αρχικώς τουλάχιστον ε, φαίνεται να είναι πιο συντονισμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και χώρες με τις οποίες ε, συνάπτονται εμπορικές συμβάσεις. Και οι εμπορικές συμφωνίες είναι ε, ένας από τους τρόπους που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να έχει πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους. Ωστόσο, η επιλογή αυτή, η επιλογή του να συνεχίσουμε ως ε, γίνονται τα πράγματα τώρα, ε, ναι μεν είναι η πιο απλή, η πιο εύκολη ε, και η πιο βολική, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν επιφέρει και αρκετά προβλήματα. Το πρώτο είναι η ενεργειακή εξάρτηση. Απλώς αλλάζουμε προμηθευτή. Αντί να εξαρτώμαστε από τη Ρωσία, εξαρτώμαστε από τις ΗΠΑ και από τον Καναδά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, αλλά η εξάρτηση εξακολουθεί να υπάρχει. Δεύτερον, η πολιτική κυριαρχία. με έδειξε να ακούσω στην αρχή τη συζήτηση ότι με τη συμφωνία TTIP μπορούμε να φτάσουμε σε ενεργειακή ασφάλεια. Και με εντυπωσίασε αυτό, διότι αν του, στην TTIP έχουμε και ενεργειακό κεφάλαιο, σε περίπτωση που υπάρχει διαμάχη μεταξύ ε, ενεργειακών κολοσσών ή χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η χωρων μελων τη ευρωπαικη ενωση αυτη η διαμαχη θα επιληθεί σε ένα διεθνέ ε, δικαστήριο που δεν έχει την ε, νομιμοποίηση που του δίνουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πολιτική κυριαρχία σε ένα θέμα ζωτική σημασία όπω είναι η ενέργεια, θα την αφήσουμε σε ένα διεθνέ δικαστήριο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ή θα το δημιουργήσουμε ή δεν θα το δημιουργήσουμε, είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, για παράδειγμα, που γνωρίζουν πολλοί από εσά, ε, περιορίστηκε ουσιαστικά και είναι απλώς κενό γράμμα, απλώς και μόνο γιατί στο τμήμα των διαπραγματεύσεων που έγινε στον Καναδά και στις Ηνωμένε Πολιτείε δεν το ήθελαν. Αυτό το οποίο ήθελε να μειώσει τις εκπομπές των καυσίμων για να τηρήσουμε την κλιματική μας δέσμευση άλλαξε λόγω των διαπραγματεύσεων. Τι θα γίνει αν αυτό γίνεται ήδη στις διαπραγματεύσεις με τη συμφωνία όταν υπεγραφεί. Στη συνέχεια υπάρχει ένα κλιματικό χάος. Αναφέρομαι σε κλιματικό χάος γιατί είναι καλύτερο ως όρος από την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν διάφορες ενεργειακές πηγές τις οποίες ακούμε πολύ συχνά, για παράδειγμα τα καύσινα, το ε, φυσικό αέριο, το φράκινγκ και άλλες πηγές. Και εδώ έχουμε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που έχουμε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα που είναι μεγαλύτερε από τα συμβατικά καύσιμα. Ε, το να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν είναι απόλυτα σωστό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρίτο καταναλωτή ε, πρωτογενού ενέργεια και αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να προσπαθεί απλώ να καθορίσει πού θα πάνε οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Διότι πολλέ από αυτέ τι πηγέ απαιτούν επενδύσει και επομένω ο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις πηγές. Η τέταρτη πηγή θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα, τα άλλες ευκαιρίες, δηλαδή το κόστος τη ευκαιρία. Όλες αυτές οι νέες πηγές ενέργειας χρειάζονται επενδύσεις. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό θα πρέπει να γίνει, γιατί αλλιώς ε, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ορεκτικά καύσιμα. Και αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πέμπτο στοιχείο, ε, αυτό το οποίο μας οδηγεί τελικά στο πιο σημαντικό, ότι φτάνουμε στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Τα ορεικτά ε, καύσιμα είναι πεπερασμένη ενέργεια και τελικώς θα βρεθούμε στο ίδιο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχω άλλα τρία λεπτά στη διάθεσή μου. Αυτό το διάγραμμα είναι το διάγραμμα της, του ανώτατου ορίου του πετρελαίου του Χούμπερτ. Ε, πρόκειται ένα μοντέλο που δείχνει το, όριο του, το ανώτατο όριο του πετρελαίου, κάτι το οποίο συζητάτε τα τελευταία χρόνια και αυτό μας δείχνει πότε θα φτάσουμε στο πικ, στην αιχμή και πότε θα αρχίσει να μειώνεται η παραγωγή. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να μειώνεται η παραγωγή πετρελαίου, τότε που θα έχουμε την κορυφή που σύμφωνα με κάποιους έχει περάσει. Κάποιοι λένε για το 2006, κάποιοι άλλοι για το 2010 ε, αλλά από το σημείο αυτό και πέρα, από το σημείο εχμέ, θα αρχίσει να μειώνεται η παραγωγή πετρελαίου. Και όλοι αυτοί οι οποίοι εξαρτώμαστε από, την, ε, από τα καύσιμα δεν θα έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Και όλες αυτές οι ενέργειες που προκύπτουν τώρα, τα μη συμβατικά πετρέλαια, ε, το σχιστολιστικό φυσικό αέριο, το φράκινγκ και όλα αυτά, είναι απλώ ένα τμήμα ε, το να συνεχίσουμε λοιπόν να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε το ίδιο μοντέλο ενεργειακής κατανάλωσης με αυτές τις πηγές ενέργειας δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Ε, απλώς θα παρατείνουμε κατά 3, 5, 10 χρόνια για να ξαναβρεθούμε στο ίδιο σημείο ε, μόνο που στο μεταξύ θα έχει επιδεινωθεί η κλιματική αλλαγή και δεν θα έχουμε αρκετούς πόρους για να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε αλλαγή μοντέλου. Αυτές ε, οι διαφάνειες, για να ολοκληρώσω, ε, άκουσα κάποια σχόλια για το πώς ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες αποκτούν ενεργειακή αυτονομία, για τις πρεβλέψεις για το σχιστολιστικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από σχιστολιστικές πηγές. Και να σας πω ότι οι τελευταίες εκθέσεις ε, και αυτή είναι μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature, καταδεικνύουν ότι τα προγνωστικά ήταν εντελώς λαθασμένα και ήταν αβάσιμα. Αν συνδυάσουμε όλα τα διαγράμματα που έχουμε από πάνω θα δείτε τις προβλέψεις και βρισκόμαστε περίπου στο ίμιση ε, βάσει πηγών της ε, ε, Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας και η πιο αισιόδοξη που είναι στα αριστερά είναι της Goldman Sachs. Περιέργως η Goldman Sachs που είναι αυτοί οι οποίοι παραποίησαν τους λογαριασμούς της Ελλάδος ε, προς το συμφέρον τους, είναι αυτοί που ε, μας λένε τώρα ότι υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο που θα μπορέσει να προκύψει από το φράκινγκ. Και το θέμα είναι ότι πίσω από αυτό το σχιστολιθικό φυσικό αέριο βρίσκεται ένα, μια, μια ακόμα χρηματοπιστωτική απάτη. Ε, θα βρεθούμε λοιπόν με μια, ενώπιον μιας ακόμα χρηματοπιστωτικής απάτης και αυτό δεν έχει κανόνι νόημα. Υπάρχει μια άλλη πρόσφατη μελέτη ενός ε, ε, γνωσμένου κύριος ε, γεωλόγου που λέει ακριβώς το ίδιο, το γαλάζιο είναι η πραγματική ποσότητα φυσικού αερίου και το κόκκινο είναι τα προγνωστικά. Και εδώ έχουμε τα ίδια προγνωστικά για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά ήταν υπερβολικά σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία και δεν θα υπάρξει τόσο πετρέλαιο και τόσο ενέργεια όσο έχουμε αυτή τη στιγμή στο μέλλον. Το θέμα λοιπόν είναι Έχω ένα λεπτάκι ακόμα, απλώς για να ολοκληρώσω, να σας πω. Ένα λεπτό, ναι, σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν και να σας πω το εξή, να τονίσω κάτι. Καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο είναι φτηνή ενέργεια και οι τιμέ είναι πολύ χαμηλέ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό είναι συγκυριακό και οφείλεται σε κερδοσκοπικά συμφέροντα και μόνον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί την αλλαγή, προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο πλαίσιο και που θα έπρεπε να βρούμε τρόπου να μειώσουμε όμω την ενεργειακή κατανάλωση, να δούμε πώ μπορούμε να έχουμε λιγότερε μεταφορέ ε, και στι πόλει μα και στη μεταφορά εμπορευμάτων ή στην βιομηχανία μα, πώ μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πώ μπορούμε να παράγουμε ανανεώσουμε πηγές ενέργειας και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα μοντέλο γεωργίας ε, οικολογικό, το οποίο ε, είναι ε, βασισμένο πολύ λιγότερο σε ορυκτά καύσιμα. Αλλιώς θα βρεθούμε σε μια, ε, στην ίδια κατάσταση, με χειρότερη κατάσταση για το περιβάλλον όμως, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και λιγότερους χρηματοοικονομικούς πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις αλλαγές που θα είναι απαραίτητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much, Mr. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν ο γύρος των συζητήσεων. Ε, είχαμε μία ώρα ανάμεσα στις 3 και τις 4 το απόγευμα. Τώρα λοιπόν μπορούν να υποβληθούν οι ερωτήσεις και εγώ ξεκινώ με μία ερώτηση προς τον κύριο Ολεχνόβιτς. Η ερώτηση μου αφορά τις εξαγωγές LNG, ε, υγροποιημένου αερίου, από τις ΗΠΑ ε, προς την Ευρώπη. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ ε, έχουν μια πιο ελκυστική αγορά και ε, πολύ πιο καλές με τις ασιατικές χώρες. Τα τερματικά θα μπορούσαν να είναι στην Κίνα ή και στην Ιαπωνία από το να είναι στην ε, κεντρική Ευρώπη. Πώς μπορείτε να το παρεμποδίσετε αυτό. Και η άλλη ερώτησή μου αφορά την πλήρη απαγόρευση του αργού πετρελαίου. Και αυτό είναι πρόβλημα για μας. Το άνοιγμα των αγορών, γιατί αυτό σημαίνει το σημαίνει άνοιγμα των αγορών. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Γκονζάλες Τεγιάντα. Η παραγωγή βιοκαυσίμων και τι είδου επιπτώσεις θα υπάρχουν από το TTIP. Όπως γνωρίζετε, τα βιοκαύσιμα δεν είναι και τόσο καλή ιδέα, κυρίως κάτω από το πρίσμα της ε, έμεσης χρήσης της γης. Προτείνω λοιπόν στα βιοκαύσιμα να υποχωρήσουμε λιγάκι από αυτήν την ιδέα. Και ερωτώ, εσείς ε, πώς βλέπετε τις επιπτώσεις της συμφωνίας TTIP στην παραγωγή βιοκαυσίμων και στη σχετική νομοθεσία ε, και θα ήθελα να δώσω και το λόγο στον αδελφό μου μας ε, να κάνει ερωτήσεις. Δεν έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια ποιες είναι οι δικές σας απαιτήσει ε, από το TTIP. Εσείς μιλήσατε για την μεταγκατάσταση των επιχειρήσεων, εσείς μιλήσατε για τον, την ενεργειακή διαδρομή, αλλά τι προβλέπετε στη συμφωνία TTIP. Δηλαδή, μήπως δεν θα πρέπει να περιορίσουμε τους δασμούς λόγω του ότι υπάρχουν ε, και διαφορετικές ε, συνθήκες ανταγωνισμού στον κόσμο ή μήπως ε, θα πρέπει να εισάγουμε έναν ειδικό κανόνα περί διοξιδίου του άνθρακα και κλίματος στη συμφωνία για το TTIP. Και όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια, ζητάμε να υπάρχει ένα ενεργειακό κεφάλαιο με βιώσιμα κριτήρια. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ζητάμε ε, μέτρα ενεργειακής επάρκειας, γιατί υπάρχει ε, συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη στο, στο θέμα της ενέργειας. Και ρωτώ ποιες είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσει μας σε αυτή τη συμφωνία TTIP. Συνάδελφος ε, Κέλλη, παρακαλώ ερώτηση ενός λεπτού. Με πολύ ενδιαφέρον σας άκουσα. Αυτά που είπατε είναι σωστά. Έχουμε την υποχρέωση να, τα, να πείσουμε τους πολίτες για όλα αυτά, να τους τα πουλήσουμε ε, και να υπάρχει θετική ανταπόκριση. Η ερώτησή μου και για τους δύο. Αν δεν συμφωνήσουμε ε, πάνω σε αυτή την ευκαιρία ε, ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, για μας όσον αφορά τη μη χρησιμοποίηση της ενέργειας ε, και των πρώτων υλών που θα μπορούσαν να μας προσφερθούν. Και κάτι άλλο. Είπατε το fracking και μπορεί να μας αρέσει και πολύ, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση. Ή να παραμείνουν και να διατηρήσουμε για όσο καιρό μπορούμε τον αγωγό από τη Ρωσία. Η κυρία Κίρτον Θα ήθελα να επανέλθω στο εξής. Με εντυπωσίασε το ότι στι διαπραγματεύσει ΤΥΠ υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι κατά την άποψή σα τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το κεφάλαιο. Γιατί από το δικό μου το πρίσμα ε, προσπαθούμε ε, να βελτιώσουμε τις ε, προδιαγραφές να διασφαλίσουμε ότι δεν υποσκάπτουμε τις προδιαγραφές. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που αφορούν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, στα πράσινα αγατά, στην ενεργειακή τεχνολογία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν πολλά ε, προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Μήπως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στο θέμα της ενεργειακής τεχνολογίας, ε, της επάρκειας, αν αυτά τα συνδέσουμε με προδιαγραφές και είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Αυτά που ακούμε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι περιορισμοί στο πετρέλαιο και το αέριο. Όμως οι εξαγωγές δεν αφορούν μόνο αυτά τα δύο προϊόντα. Τι άλλο πρέπει να περιλαμβάνει το κεφάλαιο. Ο κύριος Γκουμπάτσεκ, κοιτάξτε, ε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ολανκόβιτς ε, στη γλώσσα μου Κύριε Πρόεδρε, έχω μία ερώτηση σε αυτό που είπατε σε σχέση με το εξής. Η χημική βιομηχανία είναι πολύ σημαντική και για την κεντρική Ευρώπη. Είπατε ότι σε πέντε χρόνια αν μειωθούν οι δασμοί κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό τότε η χημική βιομηχανία στην πόλη θα έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, στο σύνολο μάλιστα της Ευρώπης, όχι μόνο στην Πολωνία. Και ε, ρωτώ, πόσο θα περιοριστεί αυτή η αγορά κατά την άποψή σας και επίσης ε, πόσες θέσεις απασχόλησης ε, θα χαθούν λόγω της έλλειψης ελκυστικότητας. Ο κύριος Σαντού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με εξέπληξε η παρέμβαση του εκπροσώπου της EEP. Είχατε πολλούς αριθμούς, πολλά αριθμητικά στοιχεία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά δεν ε, αναφέρατε τα μία, τα οικονομικά στοιχεία των, μέλων του οργανισμού, του σας που έχουν ε, επωφεληθεί από τα δικαιώματα εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα και από το σχετικό του εμπόριο. Η ArcelorMittal, για παράδειγμα, η οποία επιδοτούθηκε με τέτοια δικαιώματα και δεν απέδωσε ποτέ αυτά τα χρήματα και αντιθέτως συνέχισε να εμπορεύεται αυτά τα δικαιώματα. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα ήταν μια πολιτική η οποία βοήθησε, ε, τις βιομηχανίες εκείνες που παράγουν τεράστια ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Και οι στόχοι που έθεσε η Κομισιόν η συζήτηση για το σχιστολιστικό αέριο για παράδειγμα διαπιστώνουμε διαπιστώνουμε μάλλον, θα θέλαμε να πάμε προ την ίδια κατεύθυνση που πηγαίνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο θέμα του σχιστολιστικού αερίου ή όχι. Η κυρία Ένστ, ενστε εχω μία ερώτηση είπατε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την εξοικονόμηση και όχι την εισαγωγή ενέργειας, ε, η ερώτηση προς τον κύριο Τρεγιαντά. Και ρωτώ, τι θα κάνετε με τις ε, ενεργοφόρες βιομηχανίες, ποιες είναι ακριβώς οι προτάσεις σας. Επίσης το τι τι πρέπει να απελαμβάνει για την ενεργειακή αγορά. Να εξαιρετούν κάποια ε, θέματα, να αναδιατυπωθεί και επίσης μια άλλη βασική ερώτηση, το TTIP μπορεί να μας βοηθήσει να περιορίσουμε την ενεργειακή κατανάλωση και να στηρίξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, και το χρειαζόμαστε μήπως αυτό το TTIP, αυτή τη συμφωνία για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και πράγματι θα μας βοηθήσει η συμφωνία TTIP ε, στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ο κύριος Μόησα. Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ σύντομα ε, να επανέλθω σε μία ερώτηση που έκανε και ο πρόεδρος. Δηλαδή, ε, είναι μύθος τελικά ότι το TTIP το θα αυξήσει την ε, ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη λόγω του ότι υπάρχει διαφορά με τις τιμές στην Ασία και επίσης και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν επιβάλει κάποιε απαγορεύσει. Ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο διαπραγματεύεται η Κομισιόν. Είναι όμω σχεδόν ταμπού για του Αμερικανού. Υπήρξε εξαίρεση για τον Καναδά ε, και πριν ε, και λίγο για το Μεξικό το άλλαξαν το βαρύ πετρέλαιο με το αργό πετρέλαιο. Με πάση περιπτώσει θα καταργηθεί η απαγόρευση των Πολιτειών για το αργό πετρέλαιο. Ε, και συμφωνώ επίσης με αυτό που ελέγχει ότι η ενεργική ασφάλεια δεν έχει σχέση μόνο με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προηγουμένως... Ε, ε, θέσετε το δάκτυλο επί των τύπων των άλλων ύλων εναντίον αυτών οι οποίοι ε, και κοροϊδεύουν αυτή τη συμφωνία. Το θέμα είναι, και εδώ ε, αναφέρομαι στον κύριο Λεχνόβιτς, Εάν ε, ε, εσείς στην παρουσία σας αποδείξατε, μας δώσατε κάποια στοιχεία και αναφερθήκατε στην ανάγκη να υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κάνατε παραλληλισμό μεταξύ των εκπομπών διοξιδίου του άνθρωπου της αμερικανικής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αναφερθήκατε επίσης στο γεγονός ότι η Ευρώπη πήρε ε, μέτρα για να έχει προσιτή ενέργεια. Είπατε ότι υπάρχει και ανταλλαγή δικαιωμάτων ρηπών δωρεάν. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή εσείς, έχετε εκτιμήσει το κόστος των ετοιμάτων σας και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει το λογαριασμό κατά την άποψή σας. Ο κύριος Στοζενόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι αυτή η εμπορική συμφωνία, επαναλαμβάνω αυτή η εμπορική συμφωνία, δηλαδή το άνοιγμα μιας αγοράς, είναι μια πολύ σημαντική ε, κίνηση για την Ευρώπη. Και έχω μια ερώτηση η οποία ε, απευθύνεται στους δύο ομιλητές μας. Εάν δεν έχουμε αυτό το άνοιγμα των αγορών, τι θα ακολουθήσει. Ε, θα κλείσουμε την Ευρώπη ε, στα στενά της όρια, δηλαδή θα συνεχίσουμε με την εξάρτησή μας ε, από τη Ρωσία. Επαναλαμβάνω, αυτή η εμπορική συμφωνία ανοίγει αυτή την τεράστια αγορά η οποία ταυτόχρονα μας ε, φέρνει και νέες τεχνολογίες και άρει και τους πραγμούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ε, που έχουν ουσιαστικά περιχαρακώσει την Ευρώπη όπως γνωρίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους δύο ε, προσκεκλημένους μας τι ακριβώς θα συνέβαινε εάν δεν δεχτούμε αυτή τη συμφωνία. Γιατί νομίζω ότι η επιχειρηματολογία σας ε, ουσιαστικά αρνείται τα πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, ενώ εμείς θεωρούμε ότι το άνοιγμα της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στους ομιλητές μας ε, σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε. Δεν ξέρω με ποια σειρά. Να ξεκινήσετε εσείς κύριε Τεχάδα. Πόσο χρόνο έχω, πέντε λεπτά συνολικά για όλες τις απαντήσεις. Δεν έχετε και πολύ χρόνο. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε εδώ. Όλα βιαστικά τα κάνουμε. Microphone. Okay. Now is working. Καταρχάς, θα το έλεγα σκεφτόμενος και τους διερμηνείς, γιατί θα μιλήσω βιαστικά και τους λυπάμαι. Βιοκαύσιμα. Τα βιοκαύσιμα, πράγματα αυτό το οποίο απέδειξαν, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε ε, πρέπει να μιλάω λίγο πιο αργά από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τα βιοκαύσιμα, από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μάλλον να το πω αλλιώς, αυτό το οποίο αποδείχθηκε τα τελευταία έξι χρόνια, που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τα καύσιμα αυτά ως ε, μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, διαπίστωσε ότι δεν μειώνουν τόσο πολύ τις συνέπειες για το περιβάλλον, ιδέως ε, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και υπάρχει για παράδειγμα και το, ε, το βιοκαύσιμα μέσω σόγιας από την Ινδονησία που προσπαθούμε ε, να μειώσουμε τις εκπομπές αλλά υπάρχουν ε, συνέπειες για την αποψήλωση για παράδειγμα και κάποιες άλλες συνέπειες οι οποίες είναι χειρότερες από τα συμβατικά βιοκάψιμα. Υπάρχει βιοκαύσιμα εθανόλης, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ε, είσοδο της εθανόλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε μορφή όμως χρήση βιοκαυσίμου εξαρτάται πάρα πολύ και συνδέεται πάρα πολύ με την κατανάλωση πετρελαίου, διότι είναι ένα αγροβιομηχανικό μοντέλο και επομένως θα χρησιμοποιείται και πετρέλαιο και θα έχουμε δύο συνέπειες. Καταρχάς, η, ε, τα τρόφιμα τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι λιγότερο, γιατί πολύ μεγάλο τμήμα της παραγωγής ε, τροφίμων εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα και επίσης οι τιμές ε, των καυσίμων θα είναι υψηλότερες ε, για τα βιοκαύσιμα, επομένως δεν θα είναι και τόσο ενδιαφέροντα από πλευράς μεταφοράς, ε, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, όσον αφορά το fracking, αυτό που σας είπα εγώ στην παρουσίασή μου δεν είναι ότι ε, δίνεται μια σαφής ε, λύση. Αυτό που λέω είναι ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με την ε, παραδοσιακή μορφή χρήση ορυκτών καυσίμων, θα βρεθούμε ενώπιον της ίδιας ε, κατάστασης σε 10 χρόνια, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το να έχουμε εξάρτηση από το φράκινγκ, για παράδειγμα, και τα κάψιμα που μας δίνει αυτό, θα μας δώσει μια παράταση κάποιων ετών, αλλά θα ε, επιδεινώσει την αλλαγή του κλίματος και θα μας θέσει σε χειρότερη κατάσταση και επίσης θα διαθέτουμε λιγότερους οικονομικούς πόρους προκειμένου να αλλάξουμε την οικονομία μας. Ε, το φράκινγκ μπορεί να φαίνεται πολύ δελεαστικό αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να βελτιώσουμε την ενεργειακή η απόδοση των κτηρίων αυτή τη στιγμή για να έχουμε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και να μην εξαντληθούν οι φυσικοί μας πόροι, ε, να ε, έχουμε έτσι ε, καλύτερα οικονομικά ωφέλη και εξοικονόμηση ενέργειας από το να έχουμε μια ψευδοπαράταση 5 ετών για το φράκινγκ. Τώρα, για τη βαριά βιομηχανία με ένα εναλλακτικό ε, οικονομικό μοντέλο για τα επόμενα 5-10 χρόνια θα πρέπει να δούμε τι ρόλο έχουν να διαδραματίσουν ε, οι βαριές βιομηχανίες και επίσης θα πρέπει να δούμε και κάποιες ποσοστώσεις ενέργειας γιατί η κατανάλωση είναι καλύτερη ε, εάν η βιομηχανία βρίσκεται κοντά στο σημείο που καταναλώνει παρά να υπάρχει μετακατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που προσπαθεί να καταφέρει με τη συμφωνία TTIP και αυτό αποκαλύφθηκε και σε κάποιες ε, ε, αναρτήσεις ε, είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ουσιαστικά θα μειώσουν τους δασμούς και τους περιορισμούς που έχουν όταν θα κάνουν εξαγωγή ε, σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου. Αυτό προσπαθούν να κάνουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις και εμείς προσπαθούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους ε, που επαημένω ότι δεν θα βοηθήσουν το περιβάλλον για κανένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ή θα αλλάξει εκβάθρον ο τρόπος με τον οποίο ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για αυτές τις διαπραγματεύσεις ή δεν έχει κανένα νόημα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργεια ενέργεια έχουν μικρή πρόσβαση, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυρίως πηγαίνουν σε ηλεκτρικές πηγές ενέργειας. Είναι μια εμπορική συμφωνία η τύπη, τύπο όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε εμπορία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα όπω για παράδειγμα τη μεταφορά του. Και για να ολοκληρώσω, αυτό το οποίο σα είπα στην αρχή είναι ότι εξακολουθούμε να εξαρτώμαστε από τη Ρωσία. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει εξάρτηση από τη Ρωσία. Το πρόβλημα είναι ότι εξαρτώμαστε από ορυκτά καύσιμα. Και α είναι η Ρωσία, α είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. σω με την TTIP θα μπορούσαμε να περάσουμε στην εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα αυτή την φορά από τι Ηνωμένε Πολιτείε και λιγότερο από τη Ρωσία. Αλλά σε 5-10 χρόνια θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση και θα διαονίζεται η ίδια κατάσταση. Εγώ δεν θα προσπαθούσα να εξαρτώμαι από μία λύση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μία κοινή λύση και εμεί ω άνθρωποι βρισκόμαστε ενώπιον μια παγκόσμια και εμει ω ανθρωποι βρισκομαστε ενωπιον μίας παγκοσμια πρόκλησης και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ενεργειακό πρόβλημα και θα έπρεπε να είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν τήρησα το χρόνο μου αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ. Oh, Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι εντάξει, το χρόνο παραμείνατε. Από την πλευρά της στήρησης του χρόνου θα έλεγα ότι όλα ήταν εξαιρετικά. Κύριε Ολεχνόβιτς, 5 λεπτά, 5,5 και εσείς. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Ας ξεκινήσω με κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Προσπαθώ να έρθω στο ζήτημα της TTIP. Αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση ή όχι, μήπως είναι χάσιμο χρόνο αυτή η διαπραγμάτευση, μήπως καλύτερα να τη σταματήσουμε, μήπως ο κόσμος ο σημερινός μας ικανοποιεί με μια ατελή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με μια εξάρτηση της Ευρώπης από μια χώρα ενεργειακά και το τεράστιο πρόβλημα που αυτό μας προκαλεί Νομίζω η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι απλή. Πρέπει να ξανασκεφτούμε την εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, όχι κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους, και πώς θα επιδιώξει τη διαφοροποίηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξουμε και εμείς τη δική μας παραγωγή ενέργειας, την παραγωγή ενέργειας από την δική μας την πλευρά. Γιατί οι εταίροι μας δεν υπάρχουν εταίροι στον κόσμο με τους οποίους θα μπορούσαμε να βασιστούμε 100% σε αυτούς. Επομένως, θα πρέπει να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον τρόπο να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες που έρχονται για να είναι και εκείνη απαραίτητη σε άλλες χώρες στον κόσμο ενεργειακά. να μην βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση έναντι των ηγετικών ε, παικτών στην αγορά. Και έτσι έρχομαι και στην ερώτηση που μου θέσατε για την ασελογμητάλ. Δεν γνωρίζω ακριβώ τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης. Αλλά εμείς επιδιώκουμε μεγάλες επενδύσεις. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με ε, χρήματα, αλλά χρειάζεται και υποστήριξη. Επενδύσαμε πρόσφατα, για παράδειγμα, σε διελιστήρια υψηλότερης τεχνολογίας. Και για να, για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον ανταγωνιστικό κόσμο χρειάζεται να έχουμε σχέση και με άλλες πλευράς που σημαίνει ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς και γι' αυτό εμείς αντιμετωπίζουμε την TTIP ως γενικότερα μια συμφωνία ελευθερού εμπορίου και όχι ε, με τη στενή έννοια μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, ε, αν το ερώτημα είναι θα θέλαμε να έχουμε μια τέτοιου είδους σχέση, τέτοιου είδους συμφωνία όχι μόνο με τις ΗΠΑ και με τους άλλους, έχουμε άλλους. Ή θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια σχέση. Δεδομένου μάλιστα ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της ε, ενοποίησης των 27-28 κρατών μελών δεν έχει ακόμα προχωρήσει όσο θα θέλαμε. Άρα όταν εμείς εμφανιζόμαστε ενώπιον των άλλων, ενώπιον των άλλων εταίρων μας στον κόσμο είμαστε ε, ήδη σε θέση να εκφράζουμε με αλληλεγγύη ο ένας τον άλλο, το ένα κρατούς μέλος το άλλο, να εμφανιζόμαστε με μια φωνή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 28 κράτη-μέλη. Η ΣΥΠΗ e έχει μέλη από 11 μόλις ε, χώρες. Ωστόσο, ε, τις, πλέον, τις πιο πλούσιες, μιλάμε για τις 11 χώρες που είναι το 1 τρίτο το ΑΕΠ του συνολικό, το 1 τρίτο του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού λοιπόν περιμένουμε ότι η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον για πολλά χρόνια ακόμα, πρέπει να βρούμε με ποιον τρόπο θα βρεθεί σε πλεονεκτικότερη σχέση έναντι των υπολείπων ισχυρών της αγοράς. Έτσι βλέπουμε εμείς τα πράγματα έτσι απαντούμε στο γενικό ερώτημα και έτσι απαντούμε και στο ζήτημα της διαφοροποίησης. Εάν αποφασίσουμε, με όποιους όρους και αν αποφασίσουμε, να αγοράζουμε ενέργεια από τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Κλείσαμε λοιπόν το πρώτο πάνελ, το πρώτο μέρος αυτής της δημόσιας ακρόασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητέ για τη συμμετοχή τους σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Έχουν παραμείνει πολλά ερωτήματα ανοιχτά, προφανώς. Και βέβαια στο τέλος της ακρόασης θα έχουμε και πιο αναλυτική ε, συζήτηση και επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που διεξάγει ε, στην πράξη τις διαπραγματεύσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι μόνο θα επιτύχουμε το βέλτιστο δυνητό αποτέλεσμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ λοιπόν τους ομιλητές μας. Θα περάσω στο επόμενο πάνελ ομιλητών και δίνω και την συντονισμό της συζήτηση της Δημόσιας στον συνάδελφο του κύριο Λάγκη. Ευχαριστώ κύριε Μπιουζεκ. Με χαρά θα συντονίσω το δεύτερο μέρος της συζήτησης. Ίσως τώρα φτάνουμε στο, στην καρδιά της ε, συμφωνίας. Τι σημαίνει η TTIP για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα για, για ορισμένους ε, βιομηχανικούς κλάδους. Όπως είπα και στην αρτήρια παρέμβασή μου, η TTIP θα έπρεπε να βοηθήσει την ράχο κοκαλιά των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία Πία Ιμπαρτ από, από το ε, Ευρωπαϊκό Εταιρικό Παρατηρητήριο Corporate Europe Observatory έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τι δύο επιτροπέ του Κοινοβουλίου για την πρόσκληση. Εγώ θα ασχοληθώ με ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Το σύστημα ε, επίλυσης συγκρούσεων το οποίο προβλέπει η TTIP και θα δώσω παραδείγματα που προέρχονται από τον κλάδο της ενέργειας γιατί είναι κάτι που ε, αφορά άμεσα τις επιτροπές σας. Θα ήθελα να εξηγήσω πρώτα απ' όλα τι είναι αυτός ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών με επενδυτές, με παραδείγματα, ο μηχανισμός ISDS συγκεκριμένα. Θα σα δώσω ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιου είδου επίλυσης, είδους επίλυσης διαφορών, το παρελθόν. Θα εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στον τομέα της ενέργειας εάν συμπεριληφθεί τελικά αυτός ο μηχανισμός στη συμφωνία. Και τέλος, θα θίξω το ζήτημα των ζητημάτων, των θυμάτων που ε, θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι είναι λοιπόν αυτός ο μηχανισμός επίλυσης συγκρουσιών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Δίνει τη δυνατότητα στα, σε έναν επενδυτή σε μια ιδιωτική εταιρεία να επιλύσει μια σύγκρουση με ένα, μια διαφωνία με ένα κράτος εκτός του νομικού πλαισίου, του δικαιοδοτικού πλαισίου του κράτους αυτού μέσω μιας διαδικασίας διαιτησία, οι αποφάσεις οι οποίες μπορούν να προσβληθούν είναι αποφάσεις του Κοινοβουλίου, αποφάσεις εκτελεστική εξουσία είτε της δικαστικής εξουσία ακόμα, αποφάσεις δικαστηρίων. Τέτοιου μηχανισμού βασίζεται σε μια συμφωνία διεθνή βάσει τη οποία η αξίωση, η αιτίαση μάλλον του επενδυτή, της ιδιωτική εταιρεία είναι ότι έχουν παραβιαστεί οι όροι αυτή τη διεθνούς συνθήκη. Βλέπετε στο γράφημα αυτό πόσο έχουν αυξηθεί ραγδαία οι προσφυγές των ιδιωτικών επενδυτών έναντι τέτοιων αποφάσεων τα τελευταία χρόνια. 2014 Έχουμε πάνω από 600 τέτοιες προσφυγές κατά κρατών, πιθανότατα να είναι ακόμα περισσότερες. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι προσφυγές γίνονται με μυστικότητα και δεν είναι ακόμα ε, δημόσια γνωστές. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς οι ιδιωτικοί επενδυτές χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα, καθώς επίσης και πώς τα ε, συστήματα αυτά τα διαιτησίας έχουν την τάση να ερμηνεύουν την ομοθεσία το δίκαιο. Σε αυτό το γράφημα βλέπετε με τη μαύρη γραμμή τον αριθμό των προσφυγών κατά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρεβαία αύξηση του, ενώ η κόκκινη γραμμή είναι οι προσφυγές κατά της ε, Ενωμένων Πολιτειών, που επίσης αυξάνονται, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό, όπως βλέπετε. Συχνά συμβαίνει οι επενδυτέ από το βορρά να προσφεύγουν κατά κρατών του νότου. Και έχει γυρίσει μπούμερανγκ λοιπόν το σύστημα αυτό. Το διάγραμμα πίτας αυτό που βλέπετε, η μπλε, ε, το μπλε τομέα είναι περιπτώσεις ενέργειας. Ποδές του ενεργικού τομέα. Με κόκκινο οι περιπτώσεις εκείνες, οι προσφυγές εκείνες που αφορούν τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν τη μερίδα του Λέαντος. Ο τομέας ο ενεργειακός ε, έχει κεντρική θέση σε αυτό το σύστημα διαδυσίας. Χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα πολύ περισσότερο στον ενεργειακό τομέα από ότι σε οποιαδήποτε άλλο κλάδο της οικοδομίας. Ίσως γνωρίζετε ορισμένες από τις υποθέσεις. Μία έχει ήδη αναφερθεί. Μία προσφυγή της Vattenfall Σουηδική εταιρεία, κατά της Γερμανίας για 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ ζητά αποζημίωση γιατί την πολιτική της Γερμανίας για την πυρηνική ενέργεια. Έχει και κατά το παρελθόν ε, ε, υποβληθεί μια άλλη προσφυγή που δεν είχε τύχει μεγάλη δημοσιότητα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάλι κατά της Γερμανίας για τι περιορισμού που στο Αμβούργο είχε επιβάλει σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με άνθρακα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν τελικά τα περιβαλλοντικά πρότυπα να υποχωρήσουν. Η δεύτερη προσφυγή της Βάτενφαλ ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει. Μια άλλη υπόθεση είναι η Long ε, Pipe, μια καναδική εταιρεία η οποία έχει προσφύγει κατά του Καναδά γιατί η Long Pine ζητάει 200 ε, εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση γιατί το Quebec έχει αποφασίσει μορομερός μαρατόριο της υδρορογμάτωσης, του fracking. Μια άλλη γνωστή υπόθεση είναι η Mobile Investment, η οποία έχει προσφύγει ε, η Mobile Investment είναι φυγατρική της Exxon Mobile, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών στον κόσμο, η οποία έχει ε, και πάλι προσφύγει κατά του Καναδά και έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση του δικαιοδοτικού δικαστηρίου που τη δικαιώνει, γιατί ο Καναδάς έχει ε, επιβάλλει στις εταιρείε αυτές να επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη. Άλλη μια ενδιαφέρουσα προσφυγή. Και τέλος, άλλη μια υπόθεση η οποία έχει τέλεση δικήσει, η CMS Energy εναντίον της Αργεντινής, ήδη έχουν επιδικαστεί 133 εκατομμύρια δολάρια Ενωμένων Πολιτειών, γιατί η Αργεντινή είχε επιβάλει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ε, ε, ε ανώτατο όριο στις τιμές ε, του, της βενζίνης. Βλέπετε λοιπόν πώς αυτής αυτός ο μηχανισμός, ο παράλληλος, ο δικαιοδυτικός, επηρεάζει τον τομέα της ενέργειας. Τι θα συμβεί λοιπόν εάν συμπεριληφθεί ένας τέτοιος μηχανισμός επιλήξης συγκρούσεων, ο ISDS, στην TTIP. Ακριβώς περιπτώσεις σαν αυτές που περιέγραψα. Θα υπάρξουν προσφυγές και διατρέχουμε τον κίνδυνο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά να τύχει η να υπάρξουν προσφυγές εναντίον τους για τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ή επιση για οικονομικές αποφάσεις, όρια τα οποία ε, αποφασίζει ένα κράτος να επιβάλλει, όπως στην περίπτωση της Αργεντινής κατά την περίοδο της ε, κρίσης, ή θεμελιώδεις πολιτικές αποφάσεις όπως εκείνη της Γερμανίας ή όπως εκείνη του Κεμπέκ να ε, περιορίσει την υδρογραμμάτωση. όλες αυτές οι θεμελιώδεις πολιτικές αποφάσεις θα μπορούσαν να τύχουν να, να, να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής επενδυτικών ιδιωτών επενδυτών. Με αποτέλεσμα να κληθούν τα κράτη να πληρώσουν τεράστια ποσά, να σα ανέφερα δισεκατομμύρια δολάρια ή εκατομμύρια δολάρια που τελικά ε, τα πληρώνει ο φορολογούμενος και πηγαίνουν στις ιδιωτικές εταιρείες ως αποζημίωση. Υπάρχει επίσης και ένα άλλο ε, ε, αποτέλεσμα το γεγονός του, του εκφοβισμού. Το γεγονός ότι οι ίδιες οι κυβερνήσεις θα απόσχουν από το να λάβουν τέτοιε αποφάσει επειδή θα φοβούνται την προσφυγή. Πολύ συχνά το διαπιστώνουμε ήδη ότι οι ιδιωτικέ εταιρείε αξιοποιούν αυτό το σύστημα απειλώντα ότι θα προσφύγουν και έτσι επιτυχάνουν αυτό που θέλουν ή να αναβάλουν μια πολιτική απόφαση. Είναι λοιπόν και αυτό το πρόβλημα του αυτοπεριορισμού των κυβερνήσεων εξαιτία του φόβου που θα έχουν. Υπάρχει κάποιο όφελος από τη συμπεριλήψη αυτού του συστήματος στην τύπτη. Κανένα απολύτως. Δεν βοηθά ε, καθόλου τι ε, ιδιωτικέ επενδύσεις, δεν αυξάνει καθόλου τις ιδιωτικέ επενδύσεις, δεν αυξάνει την απασχόληση ούτε καθόλου την ποιότητα των προϊόντων. Διάβασα την έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναφέρεται επιγραμματικά, τηλεγραφικά στον μηχανισμό αυτόν, τον ISDS, αλλά αυτή η κίνδυνη είναι υπαρκτή, τους γνωρίζουμε ήδη. Υπάρχουν ήδη διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει τέτοιους κινδύνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η TTIP δεν θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης αντιθέτως. Η TTIP θα αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο που θα διατρέχουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης και η Ένωση συνολικά να αντιμετωπίσει τέτοιες προσφυγές και δεδομένων μάλλον του ε, πυκνού πλέγματος οικονομικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των εταιριών στις ΗΠΑ και των ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φανταστείτε πόσες από τις θηγατρικές των ε, εταιριών αυτών θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το σύστημα και τελικά να οδηγηθούμε σε πρόστιμα εκατομμυρίων. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθησυχάσει, έχει προσπαθήσει να καθησυχάσει πολλέ φορέ εσά του Ευρωβουλευτέ, λέγοντά σα: Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, έχουμε κάνει ανάλυση κινδύνου. Όχι. Η ανάλυση κινδύνου δεν μειώνει τον κίνδυνο ένα κράτο να αντιμετωπίσει μια τέτοια προσφυγή. Δεν μειώνει τον κίνδυνο το δικαιοδοτικό δικαστήριο τελικά, το διαιτητικό δικαστήριο τελικά να λάβει μια απόφαση απολύτω παράλογη. Καθώ επίση δεν μειώνει ούτε περιορίζει αυτό το φαινόμενο που σας περιέγραψα πριν του φόβου των ρυθμιστικών αρχών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα φοβευόμενοι τις προσφύγες. Επομένως, οι... τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να, να απαντήσουν σε αυτό το κίνημα που δημιουργείται, τους πολίτες που διαμαρτύρονται, στο κίνημα αυτό που είναι πολύ μαζικότερο από ό,τι νομίζετε. Γιατί νομίζετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες προσπαθούν να εισάγουν αυτό το σύστημα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρείες να υπονομεύουν και να προσφεύγουν κατά αποφάσεων εκλεγμένων κυβερνήσεων, κοινοβουλίων, δικαστηρίων. Γιατί νομίζετε ότι το επιδιώκουν αυτό, με ποιον τρόπο αυτό νομίζετε και μπορείτε να υποστηρίξετε ότι θα βοηθήσει το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μάριο Χούφεν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος ε, της ε, Γερμανικής Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Παρακαλώ. Αξιότιμε Μπούζεκ, ε, κύριε Λάγκε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα το ότι ως ε, πρόεδρος ε, της ε, Μεγαλύτερης Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μπορώ να σας παρουσιάσω την άποψη των επιχειρήσεων αυτών στο κοινοβούλιο σας. Η Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμφωνία αυτή παρουσιάζεται στη Γερμανία ως ένα από τα καθοριστικά θέματα των τελευταίων μηνών. Θα ήθελα λοιπόν να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι για μένα είναι πολύ σημαντική η συμπερίληψη των συμφερόντων των ΜΜΕ στις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Και αυτό ε, ισχύει όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά και αλλού ε, και προτάσω οι, μεσαία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζουν την ιδέα των ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών και στηρίζουν επίσης την περαιτέρω εμβάθυνση των ε, εμπορικών ανταλλαγών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ. Αλλά ως συνήθως ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Πρέπει λοιπόν να δούμε με κριτικό πνεύμα ποια είναι τα συμφέροντα της Ευρώπης και ποια αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά την άποψή μου ένα σημαντικός παράγον είναι η επικοινωνία με τους πολίτες πολίτες και με τις επιχειρήσεις. Γιατί όλοι ε, διαρωτώνται και εκπλήσονται για το ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν γινόταν τίποτα στην Ευρώπη. Τώρα ξαφνικά υπάρχει ολόκληρο κύμα διαμαρτυριών και τα πράγματα θα επιδεινωθούν περαιτέρω. Στη Γερμανία το 40% των επιχειρήσεων, μόνο το 40% γνωρίζουν τι είναι το TTIP. Ε, το 60% δεν ξέρουν τίποτα. Όσον αφορά τα λάθη και τις παραλήψεις της τελευταίας ε, επιτροπής, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Εδώ όμως θέλω να προσθέσω ότι η πρωτοβουλία της κυρίας Μάλστρομ ε, είναι μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Να σας πω λοιπόν από την άποψη των ΜΜΕ ε, τη δική μας άποψη που είναι πολύ επικριτική και αφορά διάφορους τομείς του TTIP. Αυτή η ρήτρα για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, αυτός ο μηχανισμός ESDS, ε, δεν αφορά μόνο τα ε, σημεία, μεμονωμένα σημεία του TTIP. Εμείς ε, θεωρούμε ότι εντάξει μπορούμε να κατανοήσουμε τις επενδύσεις και το μηχανισμό αυτό για επενδύσεις που γίνονται σε τρίτες χώρες. Αλλά μέχρι τώρα όμως ο μηχανισμός ε, έχει αναφερθεί ε, με πολύ ε, επικίνδυνες συνέπειες και το ότι αυτό συνδέεται με το TTIP καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μας εκπλήσει καθόλου. Δηλαδή υπάρχουν συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων εδώ και 50 περίπου χρόνια, παραδείγματος χάρη συμφωνίες ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ινδονησία. Όμως ε, παλαιότερα δεν ξέραμε τίποτα. Υπάρχει μια πεπατημένη ότι αποφάσεις ή ακόμα και διαδικασίες ε, δημοσιοποιούνται μόνο εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη. Αυτό εγώ δεν το εγκρίνω. Η έκφραση σκιώδης δικαιοσύνη ισχύει απόλυτα σε αυτήν την περίπτωση. Ακόμα και όσον αφορά την επιλογή των διαιτητών. Υπάρχουν ε, πολλές αρνητικές πλευρές που εμείς δεν τις δεχόμαστε. Μία μικρή ομάδα ε, διεθνών ε, ε, δικηγόρων ε, διεθνούς εμβέλειας είναι εκείνη η οποία συνεργάζεται με κυβερνήσεις για την επεξεργασία των συμβάσεων. Οι ίδιοι όμως είναι και εκείνοι οι οποίοι υπερασπίζονται τις επιχειρήσεις που προσφεύγουν κατά των κρατών. Μα κυρίες και κύριοι, πού είναι δυνατόν ε, να μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να υπερασπίζεται και τις δύο πλευρές. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όμως θα πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον ε, κάποια κίνητρα και στο ΣΥΤΑ θα ήταν δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, κατά κανόνα θα πρέπει να είναι γνωστός ο εντολέας, ε, όμως εδώ στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται κάποιο χρονικό διάστημα για να ρυθμιστεί το όλο θέμα. Επίσης, οι επενδυτές σε τρίτες χώρες δεν προστατεύονται. Αυτό όμως δεν ισχύει ούτε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να εφαρμόζει το δίκαιο, ούτε για τις ΗΠΑ ως κράτος δικαίου. Με λίγα λόγια, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα μη δημοκρατικό ιδιωτικό δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών και του οποίου αποφάσεις δεν μπορούν να εφεσιβληθούν. Στην ομολογία λοιπόν είναι σαφές ότι μπορεί κανείς να εφεσιβάλει μία απόφαση. Εδώ όμως δεν ισχύει αυτό. Ένα ιδιωτικό δικαστήριο συνεδριάζει και ε, κανείς δεν μπορεί να περάσει στην επόμενη βαθμίδα, να εφεσιβάλει μία απόφαση του δικαστηρίου. Ε, ίσως ε, σε άλλες περιπτώσεις οι αποφάσεις ε, να μην είναι τόσο σημαντικές αλλά εδώ είναι όμως και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν ληφθεί μια αρνητική απόφαση κατά 80% η επιχείρηση καταστρέφεται και αυτό δεν μπορεί να γίνει για τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Η Ellen Overy, δικηγορικό γραφείο, αυτά που σας λέω τα επιβεβαιώνει σε μια σχετική μελέτη. Έτσι λοιπόν μια τέτοια διαδικασία διατησίας διαρκεί κατά χρόνια, 4-5 χρόνια και κοστίζει για κάθε διάδικο 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μα ποια μικρή επιχείρηση μπορεί να επιτρέψει τον εαυτό της το ποσό αυτό και αν το επιτρέψει μάλιστα έχει καταστραφεί για να μην αναφέρω και το κόστος ε, το, της, δίκης που είναι 600.000 ευρώ. Τώρα, αυτή η ιδιαιτησία είναι μία από τις παγίδες ε, του TTIP. Κυρίες και κύριοι, αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία τα οποία όπως σας είπα υπερασπίζονται τόσο το κράτος και τα ίδια δικηγορικά γραφεία που γνωρίζουν τις αδυναμίες του κράτους είναι πάλι εκείνα τα οποία προσφεύγουν κατά του κράτους εκ μέρους των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Συγγνώμη, εσείς που είστε βουλευτές δεν μπορεί να διαφορείτε για μια τέτοια κατάσταση και θέλω να σας πω το εξής. Μια μεγάλη πολυεθνική, αυτά τα 5, 6, 7 εκατομμύρια τα θεωρεί ψίχουλα και πράγματι τα εκταμιεύει, τα δίνει στην νομική υπηρεσία και δεν ασχολείται περαιτέρω. Όμως η μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν μπορεί να καταβάλει ούτε καν το 1 εκατομμύριο και με το 1 εκατομμύριο έχει καταστραφεί, έχει πτωχεύσει. Έτσι λοιπόν με αυτές τις αρχές που ισχύουν από τη μία και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού βλέπουμε σύγκρουση δύο κόσμων. Η προστασία του καταναλωτή είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για σας και πολύ ευαίσθητο. Κυρίες και κύριοι γνωρίζετε όλοι σας ότι στη Γερμανία υπάρχει η αρχή της πρόληψης που σημαίνει αν έχετε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αυτό ε, το ελέγχουν οι αρμόδιοι για δυόμιση χρόνια μέχρι να μπει στην αγορά. Ο Αμερικανός μπορεί εκ των υστέρων να κινήσει τη διαδικασία. Βάζει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην αγορά και ε, το έρι μόνο αν υπάρξουν προσφυγές. Ε, στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλά σχετικά παραδείγματα που μπορώ να σας αναφέρω, αλλά κυρίες και κύριοι και σήμερα από την άποψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέλω να σας πω ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η προστασία του καταναλωτή είναι άρρηκτα συνδεμένη με το TTIP. Όλοι οι άμεσα αμπλεκόμενοι θα πρέπει με ανοιχτές διαδικασίες να πούνε ότι δεν πρέπει να θυγούν τα να φυγεί το υψηλό επίπεδο προστασίας του κατανοητή Και τελειώνοντας να πω λιγάκι για το Συμβούλιο Ρυθμιστικών Διατάξεων που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν ε, ιστορικές προδιαγραφές, οι οποίες ε, προδιαγραφές αυτές ε, είναι και προδιαγραφές που δίρκησαν, που μέχρι να θεσπιστούν χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα το να τις ανταλλάξει αυτέ αυτές ε, κανείς τις προδιαγραφές με άλλες, το TTIP, αυτό είναι παράλογο. Ούτε και πρέπει να υπάρχει ένα closed shop, ε, μια κλειστή λέσχη όπου δεν εκπροσωπούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ούτε και οι εθνικοί βουλευτές. Ούτε είναι δυνατόν η κυριαρχία των εθνικών κοινοβουλίων να φαλκιδευτεί με αυτή τη συμφωνία. Εγώ δεν ξέρω σχεδόν τίποτα για αυτό το Συμβούλιο των Κανονισμών. Υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή πρόταση, αλλά σε τελική ανάλυση οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε συμβιβασμού. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε και την πρόταση της άλλης πλευράς των Αμερικανών. Η πολιτική ρυθμίσεων δεν είναι αμεληταίο θέμα και οι καλές προθέσεις δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται και στην πράξη όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισακούνται σε, μια, σε ένα τέτοιο Συμβούλιο Ρυθμίσεων και Κανονισμών ε, στον τομέα της ε, ηλεκτροτεχνολογίας, της Ηνωμένε ε, Πολιτείες. Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει ε, χωρίς ε, κάποιες ειδικέ πλακέτες, πιστοποιήσεις. Βεβαίως αυτές δεν χορηγούνται από το κράτος, αλλά έχουν προκύψει από την πρακτική εφαρμογή. Ως εκ τούτου η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να θεσπίσει επ' αυτού και αυτή είναι μια μεγάλη παγίδα του TTIP, δηλαδή να υπάρχει μια μονομερής αναγνώριση προδιαγραφών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Γερμανίας στηρίζουν βεβαίως το να καταργηθούν οι φραγμοί στο πλαίσιο του TTIP και να υπάρχουν ε, ουσιαστικότερες εμπορικές ανταλλαγές. Αλλά αν δεν αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που σας περιέγραψα, φοβάμαι ότι το TTIP θα εξελιχθεί σε ένα αντιέξοδο, ένα στίχος πάνω στον οποίο θα πέφτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω μιλήσει με αρκετά κράτη τα οποία ε, τάσσονται με τη δική μας την πλευρά. Ε, τα κράτη αυτά θα έρθουν στις Βρυξέλλες, θα πούν τη γνώμη τους. Έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο των γερμανικών, της Γερμανικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων που έχει ακριβώς την ίδια άποψη όπως και εμείς αλλά και με τη Βέρντι, ένα μεγάλο συνδικάτο της Ευρώπης που και αυτοί λένε ότι εδώ πρέπει να προστατευτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, να δώσω το λόγο στον Λάντισλαφ Νόβακ από την χημική βιομηχανία της Τσεχίας της Τσεχικής Δημοκρατίας. Συμμετέχει φυσικά στην Ομοσπονδία και είναι και μέλος του ΣΥΒΕΚ. Έχει τον, λόγο παρακαλώ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Όπως είπατε, τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Λάγκε, κύριε Μπούζεκ. Diplomatic ε, diplomatic uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Και ε, είστε άλλωστε ένα αξιοσέβαστο τμήμα των Ευρωπαϊκών Αρχών. Uh, uh, some geopolitical... Θα μιλήσω λίγο για τη γεωπολιτική διάσταση της TTIP και μετά θα σας δώσω και κάποια στοιχεία, ε, κάποια σημαντικά θέματα, καθώς επίσης και το τι συμβαίνει στη χώρα μου, στην Τσεχία, με την TTIP. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι δεν είναι διαγωνισμός ε, εδώ Ευρώπη εναντίον του υπόλοιπου κόσμου, ούτε κάποιος εσωτερικός διαγωνισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να ξεκινήσω με την ε, ιστορική άποψη. Ιστορικά η Ευρώπη, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδά είναι ε, φυσικοί σύμμαχοι για αιώνες άλλωστε και τμήμα του πολιτισμού κατάγεται από την Ευρώπη στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, ο πληθυσμός ε, έχει τις καταβολές του εδώ. Ε, και πριν από κάποιους αιώνες αυτοί όλοι μετανάστευσαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επιπλέον, ε, οι αξίες είναι πανομοιότυπες, ε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία ε, με μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική προσέγγιση επίσης. Η διαφορά έγκυται στην αποδοχή της αρχής της πρόληψης που είναι πολύ πιο ισχυρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης στο κοινωνικό σύστημα και οι δύο κοινωνίες δημιουργούν μια βάση για τη διαπραγμάτευση προκειμένου να καταλήξουν σε μια δίκαιη συμφωνία. αυτή τη στιγμή οι ενεργειακές πηγές και οι πηγές ε, ζωοτροφών της και πρώτων υλών τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται πρωτίστως από άλλους. Ε, και αυτή τη στιγμή και από τις δύο πλευρές ε, του Ατλαντικού υπάρχει ζήτηση για μια ομαλή, ισχυρή, ισότιμη συμφωνία. Κάποια στοιχεία. Οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού δημιουργούν το 60% του ΑΕΠ παγκοσμίω. 33% του παγκοσμίου κύκλου εργασιών του εμπορίου, 30% των παγκοσμίων υπηρεσιών και όλο αυτό συνολικά ανέρχεται σε ένα δις ε, ανθρώπους, επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια δύναμη. Ε, κάποια στοιχεία από το χημικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ε, και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος σε χημικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 26 δισεκατομμύρια ε, ευρώ και οι εισαγωγές δημιουργούν περίπου 20 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ. Το πλεόνασμα λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ επιτησίως. Και αυτό φυσικά ε, υποδηλώνει και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν συναλλαγές και πολύ καλές σχέσεις ε, σε επιχειρηματικό επίπεδο. Χονδρικές εκτιμήσεις τώρα ε, εξοικονόμησης χρημάτων απλώς ε, λόγω της μείωσης ή της μεταφοράς δασμών και της εναρμόνισης των προδιαγραφών ε, και του, της σχετικής νομοθεσίας είναι της τάξης του 1,5 δις ευρώ ετησίως. Ε, πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο εξής, ε, επίσης μας λέει πολλά. Θα ήθελα να ε, περάσω τώρα στα σημαντικά ζητήματα. Κάποια από αυτά τα ανέφεραν ήδη οι προλαλήσαντες. Καταρχάς, έχουμε το θέμα της νομοθεσίας. Τα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ είναι διαφορετικά και η μηδέα αποδοχή ή ακόμα και η αμοιβαία αναγνώριση συγκεκριμένων ρυθμιστικών προτύπων στον χημικό τομέα είναι σχεδόν αδύνατη τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται. Ε, θα μπορέσουμε όμως να επιταχύνουμε την ε, αξιολόγηση για να ε, έχουμε κάποιες ρυθμιστικές απαιτήσεις πιο ομοιόμορφες και αυτό είναι το επιθυμητό. Το ουσιαστικό για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το χημικό τομέα είναι να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλε και ενέργεια και χωρίς προβλήματα. Για όλες, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να ε, μην υπάρχει χειρότερη ανταγωνιστικότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξ αρχής. Κάποια από τα κράτη-μέλη ζητούν ε, μεταβατική περίοδο για την πλήρη άρση των δασμών, κάτι το οποίο φυσικά είναι λογικό. η πρόσβαση σε γεωργικές πρωτεσίλες είναι επίσης πολύ σημαντική και ε, υπάρχει και η ψηλά αναπτυσσόμενη ε, ε, ευρωπαϊκή αγορά ε, που βασίζεται σε βιολογικά ε, προϊόντα. Προηγουμένως, αναφέρθηκε ο προλαλής σας στην μεγάλη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι το φλέγον ζήτημα, αλλά είναι πολύ πολιτικό το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα τώρα να σταθώ στα άλλα σημεία. Τι γίνεται στην τσεχική δημοκρατία ε, και στην ε, ε, χημική βιομηχανία της Τσεχίας. Θα ήθελα να σας πω ότι οι γνώσεις για την TTIP δυστυχώς ακόμα είναι περιορισμένες και δεν έχουμε και πολλά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για την TTIP, διότι αυτό φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Η TTIP ε, δεν είναι ο διάβαλος ε, όπως ε, παρουσιάζεται από κάποιους. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου τη Τσεχική Δημοκρατία έκανε μια αξιολόγηση επιπτώσεων για να δει ε, τι συνέπειε θα έχει η TTIP σε όλους του τομεί και στο χημικό τομέα. Συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία αυτής της εξ και προσπαθούμε να δούμε ε, τους όρου και τις προϋποθέσεις ε, της μελέτης. Αυτή τη στιγμή έχει δημοσιευθεί ένα τμήμα της μελέτης και κατά πάσα πιθανότητα σε δυο τρει μήνε θα έχουμε τη συνολική μελέτη. Η Ένωση Χημικών Βιομηχανών έχει ξεκινήσει και ένα εσωτερικό ερατοματολόγιο για το TTIP μεταξύ των μελών μας που αριθμούν 140. Η πλειονότητα των μελών μας είναι υπέρ της TTIP. Κάποιοι εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις, οι οποίες κυρίως σχετίζονται ε, με το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης ε, στην, ε, στις πηγές ενέργειας και ε, ο ακρογωνιαίος λίθος ε, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χωρίς καμία εξαίρεση θα είναι αυτός. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις από την TTIP και περιμένουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια ε, για τις διαπραγματεύσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια ε, για να μπορέσουμε να έχουμε ίσως κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερα στοιχεία για την TTIP. Επομένως, αυτό το οποίο θα μπορούσα να πω ε, εν είδη σύνοψης είναι ότι η προκαταρκτική άποψη της χημικής βιομηχανίας Ε, είναι ότι κυρίως υποστηρίζουμε στην τσεχική ε, δημοκρατία και στις γειτονικές χώρες η χημική βιομηχανία είναι υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης της συμφωνίας υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι τα θέματα που σχετίζονται με το κεφάλαιο της ενέργειας και των πρώτων υλών θα ε, είναι κατάλληλα ισορροπημένα. Η τσεχική δημοκρατία εν γέννη είναι υπέρ Ε, και νομίζω ότι αυτό αντανακλά και την προσέγγιση της τσεχικής χημικής βιομηχανίας. Ε, αυτό που έχει ενδιαφέρον να σας πω είναι ότι υπάρχουν φυσικά κάποιες ε, αμφισβητήσεις και μεταξύ των μελών μας, κυρίως ε, από πλευράς δηληστηρίων και πετροχημικής βιομηχανίας και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να μην υπάρχει ισόρροπη συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό στην πράξη και θα μπορούσε ίσως να μειώσει και την ανταγωνιστικότητα για κάποιες επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε επίσης και η κατάσταση ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καλή θέση, τουλάχιστον στη χώρα μας. Ε, υπάρχει μεγάλη βέβαια επιβάρυνση από την νομοθεσία, από τη χημική νομοθεσία, και επομένως η TTIP θα μπορούσε ίσως να τις βοηθήσει εάν είναι μια ισορροπημένη συμφωνία για να μπορέσουν να επεκταθούν και πέραν των συνόρων. Ε, ένα γενικό συμπέρασμα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι εμείς υποστηρίζουμε την TTIP υπό την προϋπόθεση ότι θα ε, διευκρινιστούν κάποιες ε, αμφιβολίες και θα διασκεδαστούν κάποιες ανησυχίες και φόβοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρώτα στον Πρόεδρο. Μια ερώτηση για την κυρία Έμπελχαρτ. Αυτός ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιωτικών εταιρείων και κρατών, που είναι πολύ σημαντικός, εάν δεν τον θέλουμε, ποια είναι η εναλλακτική λύση. Ένας για παράδειγμα, μηχανισμό επίλυση συγκρούσεω μεταξύ κρατών, μεταξύ κυβερνήσεων, θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε στη βιομηχανία και τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ποιο είναι ο κλάδο τη οικονομία που πιστεύετε ότι είναι ο πλέον ευαίσθητο και θα μπορούσε να πληγεί περισσότερο από την TTIP. Και μα ενδιαφέρει η απόψη σα γιατί εκπροσωπείτε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει σε μια μεγάλη χώρα κιόλα ποιοι είναι οι δυο τρει πιο ευαίσθητοι, τα τρια πιο ευαίσθητα θέματα, κέρια θέματα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε, να, τις, ε, να γνωρίζουμε τη στάση να τηρήσουμε εναντί αυτών των θεμάτων στην διαπραγμάτευση. Κύριε Νόβακ, ε, για εσά που εκπροσωπείτε τη χημική βιομηχανία, υπάρχει το πρόβλημα του κανονισμού REACH και των περιβαλλοντικών προτύπων. Πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς σε αυτά τα θέματα. μπορούμε, πιστεύετε, να διατηρήσουμε τα υψηλά πρότυπα από την Ευρώπη στη χημική βιομηχανία και να τα κρατήσουμε στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως καταφέραμε πριν από περίπου 10 χρόνια. Νομίζετε ότι γίνεται αυτό. Ο Πρόεδρος. Εγώ μια ερώτηση για τον κύριο στην έκθεση που έχω προετοιμάσει έχω ένα κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς μπορεί να αυξηθούν οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες για αυτές τις επιχειρήσεις. Εσείς τι θα θέλατε να συμπεριλάβω στο κεφάλαιο αυτό. Και τώρα δίνω το λόγο στους υπόλοιπους βουλευτές. Έχουμε ήδη 7 άτομα στον κατάλογο των ε, ομιλητών. Η κυρία Ρένα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πάντα, πράγματι αυτές οι παρουσιάσεις που ακούσαμε μπορούν να μας βοηθήσουν στις εργασίες μας. Με η παρουσίαση του κύριου Χέβεν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Σπάνια ακούμε έναν εκπρόσωπο ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχει το λόγο τη ρητορική που είχατε εσείς. Είναι σπάνιο. Το Business Europe υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ποτέ δεν το κάνει. Ποτέ δεν έχουμε ακούσει το Business Europe να εκπροσωπεί τις θέσεις που ε, υποστηρίξατε σήμερα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 90% της ευρωπαϊκής οικονομία, γι' αυτό σας ευχαριστώ για τις θέσεις που εκφράσατε. Στην πρώτη ομιλήτρια θα ήθελα να θέσω τα ερωτήματα. Ε, μιλήσατε για αυτό το μηχανισμό, τον ISDS. Γνωρίζετε ότι προβλέπεται ήδη ένα τέτοιο μηχανισμός στην ε, ΣΕΤΑ, σε μια άλλη συμφωνία, δεν θεωρείται ότι η αποδοχή αυτού του μηχανισμού σε αυτή την περίπτωση θα είναι de facto αποδοχή του μηχανισμού γενικότερα. Τώρα, έχει υπάρξει αξιολόγηση αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει δείξει ότι υπάρχουν ορισμένε χώρε οι οποίε θα ωφεληθούν, άλλε οι οποίε θα χάσουν, ορισμένοι ε, ε, κλάδοι οι οποίοι θα ωφεληθούν και άλλοι που θα χάσουν. Και ότι θα έχει αντίκτυπο η TTIP στην ενιαία εσωτερική αγορά και οι επιχειρήσει εκεί οι οποίε βασίζονται κυρίως στις εξαγωγέ προς άλλα κράτη της Ένωσης θα είναι εκείνε που θα πληγούν περισσότερο. Θα ήθελα να μάθω αν έχετε εσεί στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλλουν να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα. Τώρα για τη χημική βιομηχανία κύριε Νόβακ, ε, στο ζήτημα του κανονισμού REACH Μήπως βρήκαν οι πολυεθνικές εταιρείες του τομέα της χημικής βιομηχανίας μια ευκαιρία να επιτεθούν κατά του κανονισμού REACH που γνωρίζουμε ότι δημιουργεί προβλήματα σε αυτές χρόνια τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ τους συζητητές ε, για τις πολύ καλές ε, παρουσιάσεις τους και να πω το εξής ευθύς εξ αρχής. Εγώ θέλω να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία ε, μιας συμφωνίας ελεύθερων ανταλλαγών. Άρα είμαι θετική. Βεβαίως και ελοχεύουν κίνδυνοι. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί, έχει χαράξει κόκκινες γραμμές και τώρα προσπαθούμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τη θέση μας ως Κοινοβούλιο. Να πω κάτι για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Ε, συμφωνώ με την κριτική που ασκήθηκε σε αυτές τις ρήτρε. Εγώ για 10 χρόνια ήμουν δικηγόρος ε, σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, παρακολούθησα πολλές ε, διαιτησίες. Σωστό αυτό που είπατε. Ε, πράγματι όλα αυτά είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Εγώ λοιπόν έχω κάνει την εμπειρία ότι όσον αφορά τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης δεν χρειαζόμαστε αυτά τα διαιτητικά δικαστήρια. Και γι' αυτό ε, συμφωνώ ε, συνάδελφοι και με αυτά που είπατε εσείς στο σχέδιό σας και έχω μια ερώτηση προς εσάς γιατί άκουσα στην αρχή που είπατε ότι είστε ανοιχτός απέναντι στη συμφωνία με κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα μήπως μπορείτε να μου πείτε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορμόμενος τελικά ποιος θα υποφεληθεί από αυτή τη συμφωνία. Θέλουμε να είμαστε θετικοί υπέρ αυτής της ε, συμφωνίας. Ε, εγώ έρχομαι και έχω πολλούς ε, οπαδούς στη Βαβαρία μου λένε τι θα μας ωφελήσει. Δίνω παραδείγματα, αλλά οι περισσότεροι λένε μα οι περισσότερες εταιρείε εκπροσωπούνται ήδη στις Πολιτείες. Και όσον αφορά τους δασμούς, τελικά πού θα ωφεληθούμε. Πού βλέπετε να υπάρχουν κάποια ωφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, σε σχέση με το TTIP και αυτό με ενδιαφέρει για να μπορώ και να προωθήσω καλύτερα αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να απευθυνθώ κυρίως στους δύο ομιλητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα ε, του μηχανισμού διαιτησίας. Καταρχήν συμφωνώ με την ουσία αυτών που είπατε. Δεν πρέπει να παρακάμπτουμε ε, τα πολύ προχωρημένα ε, δικαστικά μας συστήματα προς όφελος των ιδιωτικών δικαστηρίων. Συμφωνώ με αυτό. Όμως, επειδή δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες του, της περιπτώσης CMS-GES, ε, δεν την ξέρω αυτή την υπόθεση. Αν η Αργεντινή είχε αποφασίσει να περιορίσει την τιμή του αερίου για μια εταιρεία που δραστηριοποιόταν στην αγορά της, ενώ για μια άλλη εταιρεία που δραστηριοποιόταν και αυτή δεν έλαβε τα ίδια μέτρα, αυτό είναι ε, διακριτική μεταχείριση. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Και διερωτώ με ε, κατά πόσον ε, θα μπορούσαμε να εμπιστευτούμε τα δικαστήρια της Αργεντινής όπως εμπιστευόμαστε τα δικά μας ή ε, της Βορειοαμερικής. Εντάξει, όχι ότι θέλω να τα κατηγορήσω, αλλά δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Και αυτό που υπενήσουμε είναι το εξής, ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να είναι χρήσιμος σε αυτόν τον πλανήτη και θα πρέπει να το δούμε λιγάκι προσεκτικά. Ίσως να είναι ένα εργαλείο ε, που είναι χρήσιμο, αλλά και πάλι ίσως μπορεί να μην το χρειαζόμαστε τόσο πολύ στην Ευρώπη. Κάτι άλλο που θέλω να πω σε σχέση με αυτά που είπατε κι εσείς. Πράγματι, τα πράγματα δεν είναι τέλεια και ακόμα και αν ήταν τέλεια τυπικά, ο μηχανισμός αυτός ποτέ δεν θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί πλήρως. Είναι ένας εξοδικαστικός μηχανισμός ε, διαιτησίας ε, ακόμα και αν ήταν κάτι τέλειο δεν ξέρω αν θα μου άρεσε. Πάντως όσο έχει τώρα ας πούμε στη ΣΥΤΑ ε, βελτιώθηκε σημαντικά από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν και μπορούμε να το συζητήσουμε μετά με καφέ. Ας πούμε το παράδειγμα Delaware, το τρίτη shopping ε, δεν είναι πια εφικτό. Ε, μισό λεπτό, τελειώνεται. Λοιπόν, τρεις απόψεις μπορούμε να περιορίσουμε το μηχανισμό STS στις ΜΜΕ, γιατί όχι, εκεί δεν προκαλεί ζημιά. Αν δεν λειτουργήσει, ε, τότε τους προσφέρετε το STS. Ε, thank you very much, Chair. Ε, Κύριε Σκάρικ, Κάρινς, θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου με αυτά που ακούσαμε. Χρειάζεται να έχουμε ως νομοθέτες μια ισορροπημένη παρουσίαση των πραγματικών δεδομένων, ενώ αυτό που ακούσαμε ήταν μια ιδεολογική αντίθεση στις επενδύσεις. Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου οι οποίοι ήταν παρόντες έφυγαν γιατί θεώρησαν ότι δεν έχει καμία ενημερωτική αξία αυτό το που κάνουμε τώρα εδώ αυτή η εκρόαση. είναι πράγματι ένα θέμα ITT που πρέπει να το καταλάβουμε καλά, αλλά πολλοί την παρουσιάζουν σαν να πρόκειται να χάσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή και οι δύο πλευρές πρέπει να κερδίσουν. Και το ερώτημα είναι ποιο είναι ο βέλτιστο τρόπος να φτιάξουμε ένα σύστημα τέτοιο που να προστατεύει τις επενδύσει. Δεν έχει νόημα να ακούμε ανθρώπους που έρχονται εδώ να μας πούνε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, η TTIP, είναι απαράδεκτες και θα καταστρέψουν τον κόσμο. Είναι ιδεολογικές θέσεις αυτές, οι οποίες δεν προσφέρουν κάτι, πιστεύω, στη δημόσια συζήτηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να φύγω γρήγορα να πάω σε άλλη επιτροπή, αλλά θα, πω κάποιες, θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Είμαι απογοητευμένος που στην Επιτροπή Μηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται λόγος κατά 80% για προβλήματα που έχουμε με το TTIP. Εγώ θα προτιμούσα να ε, δώσετε μεγαλύτερο θάρρος να ε, στηρίξετε αυτή τη συμφωνία TTIP και ερωτώ τελικά με την Ινδία, με την Κίνα σε θέματα εγκατάστασης εταιριών. Προχωράμε. Και μειώνονται όμως ε, τα ποσοστά της Ευρώπης, τότε στο μέλλον ποιος θα ορίζει τα βιομηχανικά πρότυπα αν δεν επεκτείνουμε την αγορά μας. Τι είναι ε, το κακό στις ελεύθερες ανταλλαγές. Εμείς δεν γιγαντωθήκαμε μέσα από αυτές. Και προς τον κύριο Χόφεν. Κοιτάξτε κύριε Χόφεν, η, τα διαιτητικά δικαστήρια είναι μια ιδέα των ΜΜΕ των γερμανικών πριν από 50 χρόνια. Τότε το είχαν ζητήσει αυτά. Και τώρα που έχουμε μία συμφωνία ας πούμε με τους Κινέζους και αυτοί διαπιστώνουν δεν υπάρχουν διαιτητικά δικαστήρια πιστεύετε ότι θα επενδύσει κανείς πια στην Κίνα αλήθεια σας λέω εγώ πολύ απογοητεύτηκα σήμερα από αυτά που άκουσα ε, και εγώ από τη δική μου την περιοχή έχω τελείως άλλα μηνύματα για τις ευκαιρίες που προσφέρει το TTIP κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες um, Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους ε, ομιλητές, κυρία Ντάρλινγκ. Ορισμένες φορές λέμε ότι είναι ιδεολογικό το πλαίσιο όταν δεν συμφωνούμε με τις ενδείξεις που μας παρουσιάζονται και για μας είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται μια ανάλυση των υποθέσεων επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με τα ενεργειακά ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για την Επιτροπή Ήτρε και δεδομένου ότι θα υπάρξει και ενεργειακό κεφάλαιο στη TTIP αν υπάρξει. Επομένως ήταν πάρα πολύ σημαντικέ αυτές οι παρουσιάσεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, επικεντρωθείτε με πάρα πολύ στην επίλυση διαφορών. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και την άποψή σας, ε, διότι ε, ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα για, τις, ε, ε, για την νομοθεσία των επιχειρήσεων και το πώς αναπτύσσεται την νομοθεσία σε βιομηχανικούς τομείς. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις επ' αυτού. Θα είναι ένα αναδυόμενο θέμα στο θεματολόγιο μας και θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας επ' αυτού. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι σαφές για μένα και για την περιφέρειά μου, διότι προέρχομαι από μια περιφέρεια που έχει πλεόνασμα εμπορίου, πολλές επιχειρήσεις εμπορεύονται με τις ΗΠΑ και ένας από τους τομείς ε, στους οποίους υπάρχει αντίληψη ότι θα μπορούσε να υπάρχει και όφελος για την DTIP είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί δεν έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες για τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, για τα ομοσπονδιακά ε, ε, καθεστώτα και το καθεστώς ε, σε κάθε πολιτεία και θα ήθελα να ξέρω τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να βοηθήσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τέλος, για τη χημική βιομηχανία. Έχω ασχοληθεί με νομοθεσία για χημικά για αρκετά χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαφορά μεταξύ του REACH και των μοντέλων που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Κορέα, στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Αυξάνεται συνεχώ όμως η χρήση του και τίνει να γίνει ένα διεθνές μοντέλο και ο ε, κανονισμός ε, για τα χημικά των ΗΠΑ, ο Τόσκα. Πώς μπορούμε να επανέλθουμε προς ε, σύγκληση, διότι φαίνεται να αποκλίνουν όλοι αυτοί οι κανονισμοί και οι νομοθεσίες. Ευχαριστώ, η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους πρώτους δύο μιλητές ε, ε, θεωρώ ότι οι, προετοιμα... προαρουσιάσεις τους βασίζονταν σε στοιχεία, ήταν συνεπείς και δεν ήταν απλώς ιδεολογικές ή πολιτικές παρεμβάσεις και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όπως και οι συνάδελφοι, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και ε, κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να υποφοληθούν από μια συμφωνία σαν την DTIP και πώς μπορούμε να προστατέψουμε τις προδιαγραφές μας όχι μόνο σε διάφορα αγαθά αλλά ε, και τα πρότυπά μας ε, για την αγορά εργασίας και τους, ε, το εργατικό δυναμικό και επίσης το κεφάλαιο για την ενέργεια όπως είπε και η συνάδελφος προηγουμένων και το τι ακριβώς θα μπορούσαμε να έχουμε στο κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζανονάτο τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, ε, με καταλάβετε ξαπίνεις γιατί είχα ζητήσει το λόγο πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους, τους ομιλητές διότι με βοήθησαν πάρα πολύ να κατανοήσω τις ανησυχίες ε, σημαντικών τομέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι πολλά από αυτά που ακούστηκαν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, όταν θα κάνουμε και τη γνωμοδότησή μας ως Επιτροπή και θα εκφράσουμε και την άποψή μας ως Κοινοβούλιο. Η γενική ε, παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι όταν μιλάμε για την TTIP θα πρέπει να πούμε τι αλλάζει σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Όχι το πώς θα θέλαμε γενικότερα τις σχέσεις μεταξύ ημών και ενός άλλου τμήματος του κόσμου των ΗΠΑ. Οι ΙΠΑ υπάρχουν, έχουν μια πολύ μεγάλη αγορά, είναι ένας πολύ μεγάλος παγκόσμιος παραγωγός, εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη και υπάρχει και η Ευρώπη, εξίσου μεγάλη αγορά που παράγει πολλά αγωθά και τα εξάγει τα προϊόντα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι ότι αυτό το αμφισβητούμε. Επομένως, όλος αυτός ο κόσμος θα πρέπει να ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο ή μας αρχεί όσο έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε. Εάν δεν μας αρκεί ως έχει, μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και αυτό γίνεται με μία συμφωνία. Και η συμφωνία αυτή λέγεται TTIP. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν ε, επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ε, ε, εντός μιας συζήτησης σαν αυτή. Παραδείγματο χάρη, όταν αναφερόμαστε στο συστολιστικό φυσικό αέριο, φαίνεται ότι βάσει αυτή τη ε, συμφωνία υποχρεούμεθα και εμεί να παράγουμε ε, συστολιστικό φυσικό αέριο. Δεν είναι έτσι. Εάν μα βολεύει, θα μπορούσαμε να το εισάγουμε. Ε, και γι' αυτό υπάρχουν και αρκετά άλλα ζητήματα. Φαντάζομαι, για παράδειγμα, ότι για τη μικρή βιομηχανία θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ενιαία προδιαγραφή και να μπορεί να εξάγει τα προϊόντα τη σε μία από τι μεγάλε ανταγωνιστικέ αγορέ και να ανταγωνίζεται με ενιαία πρότυπα αντί να πρέπει να, προ... να διαφοροποιήσει διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους γιατί σήμερα τα πρότυπα και οι προδιαγραφές δεν είναι ενιαία. Επίσης, θεωρώ ότι ακόμα και η συζήτηση για ένα διεθνή διαιτητή, αυτό το θέμα το οποίο συζητάτε ε, πολύ, θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο λογικά. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό είναι το απόλυτο κακό. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, ζητάει ο πρόεδρος θα πρέπει ε, να δούμε κατά πόσον αυτό είναι ε, ε, ουδέτερο. Για ένα λεπτό υπερβάνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό θα μιλήσω. Καταρχάς γιατί ε, ζητώ συγγνώμη δεν άκουσα τις παρουσιάσεις σας. Αυτό το οποίο με ανησυχεί εμένα για το στόχο αυτής της ακρόασης, δηλαδή οι βιομηχανικές προκλήσεις για την TTIP, είναι η ιδέα ότι όταν εξετάζουμε τη βιομηχανία στην Ευρώπη υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας ή ανισομερής κατανομής της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη. Η απλή μου λοιπόν ερώτηση είναι ε, εάν στον τομέα σας ή στις οργανώσεις σας αξιολογείτε το ε, τον αθρηστικό χαρακτήρα, τον συλλογικό χαρακτήρα. Θεωρείτε ότι η TTIP θα είναι status quo σε σχέση με την κατανομή της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη. Θα αυξήσει τις ανισότητες ή θα τις εξισορροπήσει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα λοιπόν το λόγο έχουν και πάλι ομιλητέ για περίπου τρία λεπτά. Παρακαλώ. That's a challenge. What is the alternative to... Λοιπόν, το ερώτημα είναι ποιο θα ήταν ένα αναλλατικό μηχανισμό. Να σα ρωτήσω εσά, κύριε Μπούζικ, ποιο είναι το πρόβλημα. Και σοβαρά τη θέτω αυτή την ερώτηση. Ποιο, ποια ιδιωτική επενδυτική επένδυση από τι ΗΠΑ αντιμετώπισε πρόβλημα και τον πέταξαν έξω τα δικαστήρια στις ΗΠΑ ή τα δικαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα δικαστήρια στην Ευρώπη ή στι ΗΠΑ είναι προκατηλημένα αρνητικά εναντίον των ιδιωτικών επενδύσεων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει το πρόβλημα το οποίο ισχυρίζεται ότι θα λύσει αυτό ο δικαιοδοτικό μηχανισμό. Και αν υπάρχουν ε, ε, ε, επιμέρου προβλήματα μπορούν να λυθούν με το υφιστάμενα δικαστήρια. Δικαστήρια όπω για παράδειγμα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το, το, το, το, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου επίση. Αυτός ο μηχανισμός Εάν μια, μια ιδιωτική, επενδυτικός μια ιδιωτική εταιρεία θέλει να επενδύσει σε μια χώρα, μπορεί να κάνει μια σύμβαση με αυτή τη χώρα, η οποία να προβλέπει και την επίλυση διαφορών πιο συγκεκριμένα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να δημιουργήσουμε ένα γενικό μηχανισμό έτσι, αυθαίρετο, ο οποίος θα αξιοποιείται κατά το δοκούν όπως σας περιέγραψα. Ε, αναφέρθηκε επίση το, το επιχείρημα ότι αν τον αποδεχτούμε, αποδεχτούμε ένα τέτοιο τύπο μηχανισμό στη ΣΥΤΑ, αυτομάτως θα πρέπει να τον αποδεχτούμε και στην TTIP. Αυτό δεν ισχύει. Θεωρητικά, ένας ISDS, ένας τέτοιος μηχανισμός, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην ΣΥΤΑ και όχι στην TTIP, αλλά όπως γνωρίζετε, επειδή υπάρχουν εταιρείε τη ΕΕ, τη ΗΠΑ, οι οποίε έχουν αφηγετρικά στον Καναδά, μπορούν να αξιοποιήσουν τη ΣΥΤΑ για να προσφύγουν. Κατά αποφάσεων του Καναδά. Η κριτική λοιπόν την οποία εξέφρασα την ασκεί η κοινωνία των πολιτών όχι έναντι της αλλά και έναντι της ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της επωνομαζόμενης ε, ατζέντα για μεταρρυθμίσεις της ε, Κομισιόν. Και το ερώτημα που τίθεται επίσης είναι αν εμπεριστευόμαστε δικαστικά συστήματα άλλων χωρών. Ε, δεν νομίζω υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κράτος δικαίου δεν είναι τέλειο σε όλες τις χώρες του κόσμου, ότι υπάρχουν χώρες με προβλήματα, ακόμα και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν επενδυτέ οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτό που λέμε όμω είναι ότι ο ISDS, ένα τέτοιο μηχανισμό, δεν είναι η λύση γιατί αποτελεί αφεαυτού μια παραβίαση θεμελιωδών αρχών του κράτου δικαίου, όπω για παράδειγμα την ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση υπέρ των ξένων επενδυτών, οι οποίοι είναι οι μόνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το παράλληλο δικαστικό σύστημα που δημιουργείται και ταυτόχρονα παραβιάζει την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, γιατί εδώ δεν έχουμε ανεξάρτητους δικαστές οι οποίοι αποφασίζουν, αλλά αμοιβόμενους διαιτητές. Υπάρχουν, συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι υπάρχουν προβλήματα στο κράτος δικαίου σε διάφορα κράτη του κόσμου αλλά η, η, η, λύση δεν είναι ο ISDS. Εάν υπάρχουν προβλήματα με το δικαστικό σύστημα μιας χώρας, πρέπει να το βελτιώσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε για όλους, όχι μόνο για τους ξένους επενδυτές και σίγουρα όχι δημιουργώντας ένα παράλληλο δικαστικό σύστημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ρωτήσατε σχετικά με τα πλεονεκτήματα του, της TTIP. Νομίζω ότι Όσον αφορά την TTIP, αυτό που είναι καλό είναι ότι θα υπάρξει περιορισμός ε, των ε, μη δασμολογικών ε, φραγμών και κυρίως αναφορά την πιστοποίηση και τις αδειοδοτήσεις. Ακόμα υπάρχουν πολλοί φραγμοί στις διατλαντικές μας σχέσεις. Βεβαίως άμεσα στους δασμούς δεν θα υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα γιατί και ήδη και σήμερα ο μέσος δασμός είναι περίπου 4% άρα δεν θα υπάρχουν τεράστια ωφέλη. Είπατε άλλο θετικό το Γερμανικό Ινστιτούτο Info αναφέρεται στο ότι στη Γερμανία θα υπάρξει μία αύξηση των θέσεων απασχόλησης από 45 μέχρι 100 τόσες χιλιάδες. Αλλά το ίδιο Ινστιτούτο λέει ότι στην Αμερική όμως θα υπάρξουν άλλες περίπου 1.300.000 θέσεις απασχόλησης. Αυτά τα υπέρ, τώρα τα κατά. Τα κατά είναι τα εξής τα προϊόντα υψηλής ε, τεχνολογίας έτσι κι αλλιώς με ή χωρίς ε, TTIP ε, θα συνεχίζουν να είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο. Για κάποιες τομείς όμως για τον αγροτικό τομέα αυτή η συμφωνία θα επιφέρει πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό και εκ των προτέρων πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα ζητηθούν νέες ενισχύσεις και αναφέρω το εξής παράδειγμα. Εγώ είμαι ε, στο Υπουργείο Οικονομικών πήγαμε στον κύριο Γκάμπριελ και του είπα κύριε Γκάμπριελ τι πιστεύετε ο Γερμανός ε, τρώει καλύτερα και προτιμάει τα, τις αμερικάνικες μπριζόλες ή τις γερμανικές το αμερικανικό ε, καλαμπόκι ή το γερμανικό και είπε ο κύριος Γκάμπριελ ε, τα αμερικάνικα στέικα και το αμερικάνικο καλαμπόκι και του λέω Κύριε Υπουργέ, εσείς λοιπόν θα κληθείτε να καταβάλλετε ενισχύσεις ε, στη γερμανική κτηνοτροφία και ε, γεωργία γιατί θα έχουμε λιγότερες καλλιέργειες καλαμποκιού και λιγότερη εκτροφή βοδιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιοι γραφειοκρατικοί φραγμοί δεν είναι δυνατόν να αρθούν εν μια ανοιχτή. Όσον αφορά την ηλεκτροτεχνολογία στις Ηνωμένε ε, Πολιτείες, ε, δεν υπάρχει αυτό το, αυτή η ετικέτα CA εκεί. Έχουν άλλες προδιαγραφές, γιατί αυτή η πλακέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκδίδεται από το κράτος. Βέβαια έχει επικρατήσει και έχει διαδοθεί. Άρα τι σημαίνει όμως αυτό. Δεν υπάρχουν οι ίδιες προδιαγραφές για την έκδοση αυτής της ε, πλακέτας. Και εδώ είναι μεγάλος κίνδυνος για το TTIP, δηλαδή ε, μονόπλευρη αναγνώριση προδιαγραφών. Ε, γνωρίζω να υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά, κύριε Σίτσχοφερ. Τώρα, το να έρχεται ένας ευρωβουλευτής και να λέει όλα αυτά είναι ανοησίες, θα του έλεγα για πηγαίνετε στην εκλογική σας περιφέρεια, για πηγαίνετε εκεί στις μικρομεσαίες σας επιχειρήσεις. Ε, κανείς δεν θα σας πει ότι αυτή η άποψη είναι ανοησία. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα στη Γερμανία είναι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που τις αναφέρατε κι εσείς. Και υπάρχουν και άλλα ε, πολλά παραδείγματα για διαιτητικά δικαστήρια. Ας πούμε, η Φίλιπ Μόρις στην Αυστραλία ότι έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές ε, για τα τσιγάρα. Το εκμεταλλεύεται λοιπόν αυτό η Φίλιπ Μόρις και η Φίλιπ Μόρις τι κάνει. Μέσα από το Χονγκ ε, εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Καταλήγω λοιπόν στο εξής για τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Για αυτούς υπάρχει το Handelsblatt, αυτή η εφημερίδα. Μία από τις πιο σημαντικές ε, οικονομικές εφημερίδες του κόσμου. Τι λέει το Handelsblatt. Το Handelsblatt λέει «Προσοχή Ευρώπη». Και αυτό το άρθρο θα πρέπει να το διαβάσουν όλοι διότι εκεί αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια ότι είναι παράδοξο ε, το ότι ε, τα κράτη της Ευρώπης που έχουν τα καλύτερα δικαστικά συστήματα για την προστασία της ιδιοκτησίας και παρόλα αυτά οι Ηνωμένε Πολιτείε επιμένουν να επικρατήσουν ειδικέ ρυθμίσεις για τους επενδυτές στο εξωτερικό. Θέλω λοιπόν να σας πω το κράτος το οποίο εκπροσωπείτε εσείς ε, μπορεί να υποβαθμιστεί στην αξιολόγηση και αυτό θα ήταν καταστροφικό και μοιραίο για εσάς. Τελευταίος ο ομιλητής ο κύριος Νόβακ. But not least. Uh, couple of questions to, uh, uh, to reach and SMEs. The first one was the reach and uh, Λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε τις σχέσεις με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ήθελα να τις εκφράσω σε μία φράση. Δεν είναι καλή κατάσταση, να σας πω την αλήθεια. Εμείς κάναμε τις ε, μελέτες μας στη χώρα μου και καταλήξαμε στο συμπερασμό ότι περίπου το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα σταματήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ε, ή την παραγωγή τους ή οτιδήποτε άλλο όταν θα ε, ξεκινήσει η τρίτη περίοδος καταγραφής REITs και αυτό είναι σε τρία χρόνια. Στην Ευρώπη έχουμε χιλιάδες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 96% αυτών των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ε, υπό μεγάλη απειλή. Τι γίνεται με το REACH και την κατάσταση με το TTIP ε, ε, και το θέμα που ρωτήσατε. Ε, νομίζω ότι δεν είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε από αυτά που γνωρίζω που δημιουργούν προβλήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το REACH είναι κάτι το οποίο είναι ε, καθορισμένο και δεν μπορούμε να το ξανανοίξουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να ξανασυζητηθεί. Αποτελεί κάτι σαν τη βίβλο. Δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Και ένα ακόμα παράδειγμα να σας δώσω για το REACH. Μπορεί να θυμάστε ότι υπήρχε και μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το REACH πριν από τρία χρόνια δεν κάνω λάθο. αναθεώρηση του Ρίτς, έτσι το αποκαλούσαν... και αναφερόταν στη διαφάνεια, τη γνώση των χημικών, Καθώ επίση και το πώ το αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό το Ρίτς. Και εκεί θεωρήθηκαν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εντάξει, αλλά ω προ την ανταγωνιστικότητα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το τι ακριβώ ε, σημαίνει το Ρίτς. Θα ήθελα τώρα να ολοκληρώσω με αυτή την ε, ε, φράση υποστήριξης. Πολλοί ε, ζήτησαν μεγαλύτερη υποστήριξη για το TTIP. Εγώ λοιπόν, ο Λάντισλαφ Νόβακ, ως Τσέχος και Ευρωπαίος πολίτης, θα ήθελα να πω ότι το TTIP είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να παραμείνει η Ευρώπη εντός τροχιάς και να μην χάσουμε το τρένο της ανταγωνιστικότητας. Να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε στην ανάπτυξη και στη θέση της εργασίας. Και θα πρέπει να εργαστούμε από αυτού όλοι μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Oh, uh, Clear message. Υπάρχει ένα σαφέστατο, ξεκάθαρο μήνυμα. Έχουμε και περίπου 17 λεπτά. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Yes, we, we a lot of things this uh, afternoon during the hearing, so just a, few comments. Λοιπόν, ακούσαμε πολλά πράγματα, ελάχιστα σχόλια από πλευρά μα, καταρχά ε, για τον τομέα τη ενέργεια. Ακούσαμε για παράδειγμα για την ενέργεια ότι η ενεργειακή ασφάλεια αφορά περισσότερο την πρόσβαση σε πόρους που είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε στην TTIP και το TTIP δεν μπορεί να λύσει το θέμα της ενεργειακής μας ασφάλεια. Βεβαίως, η TTIP δεν φιλοδοξεί ούτως ή άλλως να σύσει όλο το θέμα τη ενεργειακή ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να συνεισφέρει, όπω είπαμε, αλλά ε, προκειμένου ε, να αντιμετωπιστεί συνολικά ζήτημα, το, το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και πολλά άλλα μέτρα τα οποία θα απαιτηθούν και κάποια εξ αυτών θα ανακοινωθούν αύριο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει και τη δέσμη μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση που αν δεν κάνω λάθος θα παρουσιαστεί και στο Κοινοβούλιο αύριο ήδη. Ακούσαμε και από πλευράς ε, ε, ενέργειας ότι στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε πόρους μπορεί να αλλάξουμε απλώς την εξάρτηση που έχουμε ε, ε, ενώπιον του ανατολικού μας γείτονα σε εξάρτηση από τις ΗΠΑ και καλό θα ήταν να πάμε ε, προς τον τομέα της εξαφάνισης του άνθρακα από την οικονομία μας. Αυτά τα δύο δεν αποκλούν το ένα το άλλο Σίγουρα θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση από τον ε, άνθρακα στην οικονομία μας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα περιλαμβάνει ε, το θέμα της Ενεργειακής Ένωσης, αλλά θα πρέπει επίσης να κινηθούμε και προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση, κυρίως για τα ορυκτά καύσιμα, γιατί τα ορυκτά καύσιμα ε, για το εγγύς μέλλον τουλάχιστον θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη. Πρέπει να διαφοροποιηθούμε σίγουρα και η TTIP μπορεί να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίση, ακούστηκε ότι το γεγονό ότι είναι υψηλότερε τιμέ στην Ασία ε, και η δωρεάν πρόσβαση στου ε, ενεργειακού πόρου της TTIP δεν θα μας ε, ε, βοηθήσει απαραίτητα για την οικονομία. Να σα πω καταρχάς ότι η φιλοδοξία μια εμπορική συμφωνία είναι να τεθεί ένα πλαίσιο για να επιτρέψουμε στους ενδιαφερομένους να εκμεταλλευτούν αυτό το πλαίσιο. Οι διατάξει λοιπόν που θα συμπεριληφθούν στην DTIP... θα είναι χρήσιμε για του ενδιαφερομένους και το επιχειρηματία μα υπό την προπόθεση ότι θα υπάρχει δέλεαρ μέσω των τιμών. Οι τιμέ όμω κυμαίνονται ταχύτατα, αλλάζουν. Προσφάτω είδαμε πολύ υψηλέ τιμέ ε, στην ενέργεια και ε, αυτή είναι μια κατάσταση που αλλάζει ε, ήδη και η διαφοροποίηση ε, τιμών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης μειώνεται ταχύτατα και ίσως αυτό θα μπορούσε ίσως να κάνει τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις Ηνωμένε Πολιτείες πολύ Αυτά για την ενέργεια. Ε, υπήρξε πολλή συζήτηση και για τον τομέα των χημικών. Θα ήθελα να σας διευκρινίσω λίγο την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ανέκαθεν λέγαμε ότι δεν επιθυμούμε να συζητήσουμε το επίπεδο προστασίας που αποφασίζεται και παρέχεται μέσω του ΡΙΤΣ. Εμείς κάνουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε στα πλαίσια του δικού μας κανονισμού ΡΙΤΣ. Ε, ο στόχος της διαπραγμάτευσης δεν είναι να υπάρχει πλήρη σύγκληση, γιατί τα... Ε, ε, συστήματα αυτά ε, διαφέρουν πολύ μεταξύ των, επομένως θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, ρυθμιστικών αρχών εντός των δύο συστημάτων. Αυτός είναι ο στόχος για το REACH. Ακούστηκαν πολλά για το σύστημα επίλυσης διαφορών, το ISDS, και εδώ θα ήθελα να επαναλάβω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις εν εξελίξη αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της TTIP. Ε, νέα προσέγγιση για την προστασία των επενδύσεων και του συστήματος επίλυσης διαφορών, ε, το οποίο θα τηρεί πλήρως ε, τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε έγινε μια δημόσια διαβούλευση για την προστασία των επενδύσεων και το ISDS. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα και επί τη βάση των απαντήσεων που λάβαμε έχουμε εντοπίσει τέσσερις τομείς συγκεκριμένα που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαρευνήσουμε περαιτέρω. Υπάρχει το θέμα της προστασίας του δικαιώματος να νομοθετεί κανείς, ε, την ε, δημιουργία και λειτουργία των ε, διαιτητικών δικαστηρίων, τη συνεργασία με τον, μεταξύ των δικαστικών συστημάτων και του συστήματος επίλυσης διαφορών και η διαδικασία έφεσης αυτών των αποφάσεων των διαιτητικών δικαστηρίων. Θα πρέπει τώρα να διαβουλευτούμε με τους ενδιαφερομένους, ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτούς τους τέσσερις τομείς, ως τμήμα μιας ευρύτερης συζήτησης για την προστασία των επενδυτών και ε, του συστήματος επίλυσης διαφορών, το οποίο θα ε, δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει πλήρεις προτάσεις για τις διαπραγματεύσεις για το TTIP πριν από το καλοκαίρι. Και τέλος, επειδή ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, επιτρέψτε μου κύριε ε, Πρόεδρε να πω δύο λόγια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς ορισμένες φορές θεωρούμε ότι δεν συμμετέχουν επαρκώς στις ε, εξαγωγές, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 81% των εξαγωγέων μας, 81% των επιχειρήσεων που εξάγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτές ε, οι 600.000 επιχειρήσεις και οι εξαγωγές τους αντιπροσωπεύουν περίπου το 1 τρίτο των συνολικών εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ήδη συμμετέχουν αρκετά, αλλά βεβαίως θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να συμμετέχουν ε, ε στο διεθνές εμπόριο και στο συγκεκριμένο εμπόριο με τις ΗΠΑ. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε και χαιρόμαστε που ε, αναφερθήκατε στην ιδέα ε, του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Αυτή είναι και η κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι η μόνη, η πρώτη εμπορική συμφωνία στην οποία θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε ουσιαστικά τα πάντα μεταξύ τους. Διότι ε, όλες οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία θα είναι υποφελείς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μέσω αυτού του κεφαλαίου και του μηχανισμού που θα παρέχεται στο κεφάλαιο αυτό, θα είναι πολύ πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις αυτές να εκμεταλλευτούν όλες αυτές τις διαφορετικές διατάξεις. Για παράδειγμα, εάν καταφέρουμε να έχουμε μια επιτροπή για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σίγουρα αυτό θα βοηθήσει. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, το πρώτο βήμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι να γνωρίζουν ε, μέσω πληροφοριών ποιες είναι οι συνθήκες της αγοράς και εμείς στις διαπραγματεύσεις προσπαθούμε οι δικές μας οι επιχειρήσεις και φυσικά οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ να λαμβάνουν πληροφορίες για τις αντίστοιχες αγορές και αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζουμε ιδιαίτερα στους Αμερικανούς εταίρους μας. Ε, συγγνώμη που μίλησα για περίπου 8 λεπτά, αλλά θεώρησα ότι ήταν πολύ σημαντικό για την Επιτροπή σας να γνωρίζει και την προσέγγιση μας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ και τα μέλη του δεύτερου πάνελ ομιλητών. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι παρεμβάσει σα, παρουσιάσει σα. Θα λάβουμε υπόψη τι απόψει που ακούστηκαν στι μελλοντικέ μα διαβουλεύσει, συζητήσει, εργασίε εν ώψη και τη Ολομέλεια του Μαΐου. Κύριε Μπούζακ. Κλείνοντας τη συζήτηση, θα πω ότι η συζήτηση αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική. Ακόμα και αν δεν καταφέραμε να βρούμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ετέθησαν πάντως, θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, γιατί γνωρίζουμε ότι τα θέματα είναι σημαντικά, η πληροφορική, η ενέργεια, οι μικρές επιχειρήσεις, η, η πολιτική για τη βιομηχανία, η τεχνική εναρμόνιση και ομογενοποίηση κτλ. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικά για την οικονομία της Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Υπήρου συνολικά. Αλλά Ένα ερώτημα είναι οι λεπτομέρειε. Ένα άλλο ερώτημα που ίσω θα έπρεπε να συζητήσουμε είναι οι ιδεολογικέ ερωτήσει. Γιατί και τα ιδεολογικά ερωτήματα είναι πολύ σημαντικά και απασχολούν του Ευρωπαίου πολίτε. Ίσως να έπρεπε μια τέτοια συζήτηση μάλιστα να ξεκινήσει από τα κράτη-μέλη. Τοπικά. Κατά την άποψή μου, μια τελική συμφωνία θα πρέπει να λάβει υπόψη τη τι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εν τέλει η συμφωνία θα επικυρωθεί με ψηφοφορία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαφορετικά, εάν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγνοήσει τις συστάσεις και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, υπάρχει ο κίνδυνος της καταψήφισης της συμφωνίας και αυτό θα ήταν πολύ κρίμα, μεγάλο πρόβλημα, κρίμα, θα δημιουργούσε και προβλήματα στην Ευρώπη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην κοινωνία, στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εν τέλει αυτή η απόφαση θα είναι πολιτική. Ευχαριστώ πολύ, κλείνουμε εδώ την ακρόαση. Καλό απόγευμα.